Ladies and gentlemen, good morning. Please take your seats. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Καθίστε. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πολύ ενδιαφέρουσα ημερήσια διάταξη. Καταρχάς, να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και έχουμε διερμηνία στις γλώσσες των τακτικών μελών έγκριση της ημερήσιας διάταξης Εάν δεν έχετε παρατηρήσεις, θεωρώ ότι είναι κρίθη. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα, χάρη στην καλή θέληση των πολιτικών ομάδων, θα έχουμε την συνεδρίαση για την παρουσία των ε, ε, Ρώσων στην ε, περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας. Ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες και να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα θα αναλάβει την Προεδρία για ένα θέμα ο κύριος Στέτινα. Γιατί έχω άλλες υποχρεώσεις. Να περάσουμε απευθείας στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με χαρά καλωσορίζω τους διακεκριμένους ομιλητές μας Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο από το Ισλαμικό κράτος στο Λίβανο. Θα μιλήσουμε για το ρόλο των πολιτοφυλακών. Έχουμε εδώ μαζί μας την καθηγήτρια κυρία Ελένα Αούνα. Ορισμένοι τη γνωρίζετε. Όλοι τη γνωρίζετε. Όλοι όσοι γνωρίζετε την κατάσταση στο Λίβανο γνωρίζετε και την κυρία Αούν και γενικά ως επώνυμο είναι πολύ γνωστό στο Λίβανο. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν και ο δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Τζον Γκάτς Ράτσα που είναι τμήματάρχης ε, στο τμήμα καταπολέμησης τρομοκρατίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη Μέση Ανατολή, της οποίας ο Λίβανος είναι σημαντικό τμήμα. που ήταν ε, ζωτικής σημασίας ε, εδώ και πολλά χρόνια για την ε, ασφάλεια της περιοχής. Και ε, ανεφετέρου να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια κυρία Αουν και μετά θα πάρει το λόγο και ο κύριος Τζον Γκάτ Ράτσα. Okay. So, greetings all. Ε, χαίρετε, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που έλαβα για να εξετάσουμε τον ρόλο των πολιτοφυλακών στην καταπολέμηση του ISIS. Είναι δύσκολο θέμα και δεν μπορούμε να τα βλέπουμε ε, χωρίς αποχρώσεις. Δεν είναι όλα μαύρα ή άσπρα. Ελπίζω λοιπόν ε, όλα αυτά που θα σας πω να σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς έχουν τα πράγματα και ποια είναι τα διακυβεύματα. Ποιο είναι το βασικό μου επιχείρημα. It's okay. It's all... But I didn't manage to. So, thank you. Um, So start with my core Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μου επιχείρημα. Ορισμένες ε, πολιτοφυλακές στο Λίβανο, κυρίως το Hezbollah, παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του ISIS στο Λίβανο. Αλλά η παρουσία τους και η δράση τους συμβάλλουν στην διαιώνιση ενός γενικότερου κλίματος που ε, τροφοδοτεί το τζιχαντισμό και κινήματα σαν το ISIS. Άρα οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμότητά τους βράχει πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα υπάρχουν αρνητικά, αρνητικές παρενέργειες. Για να τα καταλάβουμε αυτά, να δούμε διάφορες πλευρές. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε μια επισκόπηση των πολιτοφυλακών, μετά ποιος είναι ο ρόλος του Χίσμολα, μετά θα ασχοληθώ με τις άλλες πολιτοφυλακές και και ίσως ε, να σας εκπλήξω ότι θα ασχοληθώ και με τις ε, ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και θα καταλήξω για το πώς οι δράσεις όλων αυτών βοηθούν την επιχειρηματολογία του ριζοσπαστικού, εξτραμιστικού τζιχαντισμού. Λοιπόν, οι πολιτοφυλακές στο Λίβανο, όπως ξέρετε, στο Λίβανο δεν είχαμε ποτέ ένα βασικό στοιχείο ενός σύγχρονου κράτους δηλαδή να έχει το μονοπόλιο στην νόμιμη χρήση βίας. Και αυτές οι πολιτοφυλακές ήταν πάντα στη σκακέρα της ε, λιβανέζικης πολιτικής ζωής κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν ένας ε, απίστευτος αριθμός πολιτοφυλακών παρών και ήταν ε, διαφορετικές οι πορείες τους, οι στόχοι τους, οι συμμαχίες που σύλληπταν κτλ. Και όπως θα ξέρετε, η συμφωνία του ΤΑΙΦ που ήταν η κατάληξη του εμφυλίου πολέμου, πολέμου στο Λίβανο προέβλεπε τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών αλλά το αποτέλεσμα της εφαρμογής του ήταν άνισο. Ο Νότιος Λίβανος παρέμεινε υπό τον έλεγχο του Ισραήλ με τον στρατό του Νοτιού Λιβάνου που λεγόταν μια πολιτοφυλακή που δρούσε υπό τις εντολές του. Ο Συριακός στρατός και το Συριακό καθεστώς είχαν συμφέρον να επιτρέψουν σε ορισμένε ομάδε να διατηρήσουν ε, τον οπλισμό τους και κυρίω ωφελήθηκε το Χεσμολά που έγινε ε, ο κύριο φορέας της αντίσταση στην ε, Ισραηλινή κατοχή και τις προσπάθειες που έκανε να επηρεάσει το Ισραήλ την κατάσταση στο Λίβανο. Οι άλλοι οποίοι ωφελήθηκαν από την ηγεμονική θέση της Συρίας ήταν διάφορες Παλαιστινιακές ομάδες και ο Λιβανέζικος στρατός απλώς έλεγχε τα σημεία εσόδου σε διάφορους καταβλισμούς και αφαιρούσε το βαρύ οπλισμό. Και μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι η σταδιακή άνοδος των τζιχαντιστικών ομάδων που ξεκίνησε στη δεκαετία του 90 και αυξήθηκε πολύ στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Τώρα ποιος είναι ο ρόλος του Εσμπολά. Ο Εσμπολά είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ISIS και αναφίβολα παίζει ρόλο κλειδί στην ε, στρατιωτική αντιμετώπιση και περιορισμό των ριζοσπαστικών ομάδων. Και ο ρόλος έχει πολλές πλευρές, αυτός ο ρόλος του Χεσμολά. Πρώτα απ' όλα, το Χεσμολά έχει πολύ στενές σχέσεις από την αρχή με το Ιράν και τη Σύρια και αυτό έκανε το Χεσμολά να καταπολεμήσει τους ε, αντικαθεστωτικούς στο, στο, στη Συρία. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές προσπάθειες του, του Χεσμολά είχε στόχο την προστασία των ε, χωριών Σία και διαφόρων ε, θρησκευτικών μνημείων κοντά στα σύνορα Συρίας Λιβάνου. Παρά λοιπόν το ότι το Χεσμολά προσπάθησε να αποσυνδέσει την Συριακή με τη Λιβανέζικη πολιτική, διάφορες ε, ομάδες άρχισαν να κάνουν ε, διάφορες ε, επιθέσεις αυτοκτονίας και βομβιστικές ενέργειες με παγιδεμένα αυτοκίνητα σε σιητικές γειτονιές στο Λίβανο. Και το Χεσμολά ε, ανταποκρίθηκε με σχετικά αποτελεσματικό πρώτο, τρόπο. Συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα αύξησε την παρουσία των δυνάμεών του στην Συρία, πολεμώντας το πλάι του καθεστώτος και αυτό το αναγνωρίζουν και ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες όπως η Ρωσία και πρόσφατο ο ο Γάλλος πολιτικός. Δεύτερον, το Χεσμολάμ έχει σημαντική στρατιωτική παρουσία σε διάφορα λιβανεζικά ε, σημεία έντασης ε, στο βορρά της χώρας για να περιορίσει την επέκταση των ε, ακραίων ομάδων. Και επίσης έχει κινητοποιήσει μια σειρά από δυνατότητες ασφάλειας και συλλογής προφοριών που ανέπτυξε από την περίοδο, από την περίοδο του 90 και του 2000 σε συνεργασία με τις λιβανεζικές μυστικές υπηρεσίες. Και, τελευταίο αλλά σημαντικό, έχει βοηθήσει στην ίδρυση διαφόρων πολιτοφυλακών που πολεμούν το ISIS. μπορείτε να δείτε καταρχάς εδώ ένα χάρτη όπου φαίνεται η έκταση και οι περιοχές όπου δρά ο Χεσμπολά. Εδώ βλέπετε και ποιες περιοχές ελέγχει το ISIS που επιτίθεται και όπως είπα οι περισσότερες επιθέσεις ε, επιθέσεις του ISIS δηλαδή απευθύνονται κατά περιοχών και σημείων που ελέγχει το Χεσμολά. Βέβαια αυτός ο χάρτης δεν ε, δίνει πλήρη εικόνα. Κάποιες παρατηρήσεις. Ναι, μεν το ISIS ε, ελέγχει όλο και περισσότερο ορισμένε περιοχέ, αλλά δεν είναι η μόνη τζιχαντιστική ομάδα στο Λίβανο. Δεύτερον, οι πυρήνε τζιχάντι ε, έχουν βάση και στους παλαιστινιακούς ιδιαίτερα στο Αϊν Αλχέλουι, στο Νότο. Αλλά δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Τρίτον, σύμφωνα με έναν ε, Λιβανέζο υπεύθυνο 20.000 τζιχάντις ε, έχουν διεισδύσει στους καταβλισμούς προσφύγων στο Λίβανο όπως βλέπετε εδώ στο χάρτη σχεδόν παντού αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι η απειλή μπορεί να είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι λένε οι πηγές μας στον τρίτο χάρτη εδώ που μας τον έστειλε μια πηγή που είναι κατά του Χεσμολά αλλά μας δίνει μια εικόνα για την παρουσία του Χεσμολά και την δράση του κατά τον τζιχάντη στο Λίβανο, κυρίως στο Βορρά και την Ανατολή. Αλλά τα στοιχεία είναι από το Μάιο του 2015. Έκτοτε έχει αυξηθεί περαιτέρω η παρουσία του Χεσμολά. Ποιες άλλες τώρα πολιτοφυλακές υπάρχουν που δεν μπορούν να συγκριθούν με τον Χεσμολά αλλά θα αναφέρω ορισμένες. Το πρώτο, η πρώτη ομάδα πολιτοφυλακών ε, σχετίζεται με την προσπάθεια του Χεσμολά κατά των εξωτικών ομάδων. Ορισμένες ε, τοπικές σε διάφορες περιοχές ε, ένοπλες ομάδες έχουν ιδρυθεί κυρίως στην βορειοανατολική περιφέρεια και οι σχέσεις τους με το Χεσμολά είναι προς το παρόν άτυπες. Αλλά να σας δώσω μερικά παραδείγματα στην περιοχή στο χωριό Γαράστον Αλμπακ, που είναι χριστιανικό χωριό, δημιουργήθηκε μια ομάδα αυτοάμυνας με τη στήριξη του Hezbollah. Επίσης κατάφερε να κινητοποιήσει το Hezbollah και διάφορες ε, ομάδες που ασχολούνται με το λαθρεμπόρο ναρκωτικών, που είναι ήδη ένοπλες και τώρα ε, μάχονται και, και εκείνες οι ομάδες στο ISIS. Και από ό,τι ακούμε, Ε, μαθαίνουμε ότι το Χεσμολά στον Ανατολικό Λίβανο στρατολογεί νέους εκπαιδευμένους και ένοπλους άνδρες που δεν σχετίζονται ε, κατά ανάγκη, δεν είναι κατά ανάγκη ενσία. Και με αυτόν τον τρόπο σε ορισμένε περιοχές αντιμετωπίζουν το ISIS. Ε, κάτι άλλο που είναι λιγότερο εμφανές, το δεύτερο σύνολο πολιτοφυλακών, σχετίζονται με παλαιστινιακές ομάδες που και αυτές ομάδου, ε, συγγνώμη, και αυτές περιορίζουν τη δράση του ISIS σε διάφορους καταβλισμούς στο Λίβανο, ιδίως στο Άιν Αλχάουι. Οι Λιβανέζικες αρχές, όπως σας είπα, δεν ελέγχουν τους καταβλισμούς αυτούς. Αλλά αυτοί οι καταβλισμοί ε, είναι πραγματικές θερμοκοιτίδες για τους τζιχάντι. Και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες ε, χαμηλού επίπεδου ε, σειράξεις και συγκρούσεις σε, διάφορα, σε διάφορους καταβλισμούς, αλλά οι επιτροπές διοίκησης των καταβλισμών έχουν καταφέρει να περιορίσουν αυτές τις συγκρούσεις με συνεργασία με τις ε, ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Οπότε, να αναφερθώ τώρα στον ε, Λιβανέζικο στρατό. Γιατί τον περιλαμβάνω. Δεν είναι πολιτοφυλακή. Είναι τακτικό στρατός. Αλλά θεωρείται ότι όλο και περισσότερο ε, δράει υπέρ κάποιον και κατά κάποιον, γιατί συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό με το Χεσμολά. Προς το παρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εκτιμήσουμε το βαθμό συνεργασίας μεταξύ του στρατού του Λιβάνου και του Χεσμολά, αλλά αυτή η συνεργασία βέβαια δημιουργεί σύγχυση ως το ποιος είναι ποιος, τουλάχιστον για ορισμένους στο Λιβάνο. Σε στρατιωτικό επίπεδο το Hezbollah στηρίζει τον στρατό στις περισσότερες συγκρούσεις του με διάφορες ε, ομάδες. Είναι βέβαια το Χεσμολά καλύτερα εκπαιδευμένο και πιο έμπειρο από το στρατό του Λιβάν. Και ναι μεν προσπαθεί να είναι δεκριτική η παρουσία του Χεσμολά, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο. Όταν άρχισαν ε, οι τζιχάντες να επιτίθενται στις ε, κοινότητες ΣΥΑ, τότε ο στρατός ε, εποφελήθηκε από τη βοήθεια των δυνάμεων προφοριών, των υπηρεσιών προφοριών, του Χεσμολά και αυτό οπωσδήποτε αύξησε την αποτελεσματικότητά του. Να σας δείξω και πάλι ένα χάρτη, τον οποίο ε, επεξεργάστηκα. Για να δούμε πώς ε, ο στρατός και το Χεσμολά περιόρισαν τον τζιχάδι. Στον Νότο, αν δείτε εδώ το κόκκινο κύκλο, βλέπετε ότι ο στρατός κατάφερε να αντιμετωπίσει τον ριζοσπαστικό Σεϊχη Αχμαντ και συνεργάζεται με τις Παλαιστινιακές ε, δυνάμεις ασφαλείας στο Αϊναλ Χελουέ. Και το Χεσμπολά ε, θεωρούμε ότι συνεργάζεται πολύ στενά, αλλά με κάπως αφανή τρόπο. Δεύτερον, στο βορρά. Ο στρατός ε, παρακολουθεί το στρατόπεδο των Παλαιστινίων Άχελ Μπάρεντ όπου έγιναν συγκρούσεις με την ε, ακραία ομάδα Φάτελ Ισλάμ και επίσης είχε αναπτύξει δυνάμεις και στην Τρίπολη που είναι η μεγαλύτερη πόλη του Βορρά όπου είχαμε μια σειρά από συγκρούσεις μεταξύ Σούνι και Αλαουί ομάδων. Το Χεσμολά δεν έχει μεγάλη παρουσία στην περιοχή άρα δεν έχει και άμεση συμμετοχή. Αλλά η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική στην βορειοανατολική περιοχή τη χώρα, όπου και ο στρατό και το Χεσμολά έχουν αναπτύξει τι δυνάμει του. Και ναι, μεν προσπαθεί με διακριτικό τρόπο το Χεσμολά να στηρίξει το στρατό, αλλά το Χεσμολά θεωρείται ότι είναι ο πιο αποτελεσματικό μαχητή στην περιοχή. Και τέλο, υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο υπηρεσιών ασφαλεία, ουσιώδη και στη Βηρητό, όπου ο στρατό χρειάστηκε να αναπτυχθεί για να σταματήσει τι επιθέσει κατά των ε, νοτίων περιοχών της Βηρητού όπου είναι η Σία με πολύ σχεδή βοήθεια από το Χεσμολά. Βλέπετε εδώ παραδείγματα στο χάρτη. Αυτή η συνεργασία λοιπόν είναι πολύ αποτελεσματική. Βέβαια δεν ε, απέφυγε όλες τις επιθέσεις, δεν ε, εκρίζωσε την απειλή από τους τζιχάντι, αλλά πολλές επιθέσεις αντιμετωπίστηκαν και ε, εμποδίστηκαν εκατοντάδες τζιχάντι. Καταλήγοντας, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής ο ρόλος των πολιτοφυλακών και ιδιαίτερα του Hezbollah έχουν υπάρξει, ο ρόλος αυτός είναι αποφασιστικός για τον περιορισμό των ε, ακραίων ομάδων. Όμως ε, η παρουσία του Hezbollah στη Συρία και στο Λίβανο ενισχύει την προπαγάνδα του, των Σούνι που προπαγανδίζουν ότι ε, είναι κοινότητα που καταπιέζεται και ε, αντιμετωπίζει κίνδυνο ακόμη και εξάλληψης από τις δυνάμεις των ΣΥΑ. Και αυτή η προπαγάνδα έχει ριζοσπαστικοποιήσει πολλούς Σουνίτες του Λιβάνου. Και αυτό συνδέεται επίσης και με την πόλωση που υπάρχει στον Λίβανο και τον ευρύτερο ανταγωνισμό ε, που υπάρχει και με την Σαουδική Αραβία και το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η δραστηριότητα του Χεσμολά μπορεί στην ουσία να στρατολογήσει περισσότερους ε, τζιχάντι. Όσο περισσότερο χάνουν τις δυνάμεις τους στη Συρία και το Ιράκ ε, οι τζιχάντι και χρειάζεται να διαφύγουν. Η στενή συνεργασία μεταξύ του στρατού και του Χεσμολά μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα, διότι ο στρατός μπορεί να θεωρηθεί όλο και λιγότερο ουδέτερος και να θεωρηθεί από τις κοινότητες των Σούνι ότι δράει εναντίον τους. Ακόμη και στις ε, ε, λιγότερο ζωσπαστικές ε, ομάδες στο Λίβανο, ο ρόλος του στρατού θεωρείται αρνητικός σε πολλές περιπτώσεις στην καταπολέμηση των οπαδών του Ασύρ στην Σιδώνα, στην αντιμετώπιση της ασφάλειας στην Τρίπολη, στον Άχαρ Μπάρεντ, όπου πολλοί τζιχάντις συλλαμβάνονται, κρατούνται και σε ορισμένε περιπτώσει βασανίζονται. Ένα τελευταίο στοιχείο έχει να κάνει με την, τον εξοπλισμό διαφόρων ομάδων ε, αυτοάμυνας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον στη συνοχή του Λιβάνου. Τα όπλα, όπως όλοι ξέρετε, πιο εύκολα είναι εύκολο να τα διανύμεις παρά να τα πάρεις πίσω και είναι πιο εύκολο να κινητοποιήσεις ε, κάποιες κοινότητες παρά μετά να τις ε, αφοπλήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ και με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάτ Ράδερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με χαρά βρίσκομαι εδώ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Λίβανος είναι βασικός εταίρος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μαζί με κάποιες άλλες ε, χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Λίβανος, λόγω της ε, εφραστότητας, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω των ε, συγκρούσεων στην περιοχή, παρόλα αυτά κατάφερε να αντισταθεί στην απειλή του Ισλαμικού κράτους. Πήγαμε στην Βηρητό τον Ιανουάριο, μια αποστολή υψηλού επίπεδου, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και της Γενικής Διεύθυνσης HOME, για να συζητήσουμε την εταιρική μας σχέση με τους Λιβανέζους εταίρους μας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να ε, αντισταθούν στις σημαντικές πιέσεις που δέχονται από το ISIS και από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι η εντύπωσή μου είναι ότι παρά την εύστραστη ε, πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, ε, οι διαμάχες μεταξύ Σαουδαράβων και Ιρανών, οι θρησκευτικές ε, εντάσεις εντός της χώρας, παρά το γεγονός ότι γειτονεύει με τη Συρία, παρά λοιπόν όλες αυτές τις πολύ μεγάλες δυσκολίες, ο Λίβανος έχει καταφέρει να αντισταθεί στις πολύ ισχυρέ εξωτερικές πιέσεις. Σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με τις διάφορες υπηρεσίες και τις αρχές της χώρας, ε, εμένα με εντυπωσίασε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι στο Λίβανο, αυτό που λένε ε, με τον τρόπο που καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτος, με τον τρόπο που ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των ε, διαφόρων υπηρεσιών και αρχών, γιατί και αυτό δεν είναι πάντοτε ε, αυτονόητο. Εδώ, εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στο Λίβανο, παρά το γεγονός ότι διάφορες υπηρεσίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο διαφόρων κοινοτήτων, καταφέρνουν να συντονίζουν τη δράση τους προκειμένου να καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτος και άλλες τρομοκρατικές ομάδες. Και η δική μας δουλειά, ο δικός μας στόχος είναι πώς μπορούμε να παρέχουμε ε, βοήθεια προς τη χώρα αυτή. Συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και της ε, Τινησίας και της Ιορδανίας. Συζητήσαμε λοιπόν για μια στρατηγική αντιτρομοκρατία για το πώ θα μπορούσαμε να του βοηθήσουμε όσον αφορά την επιβολή του νόμου, την καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας, τη διαχείριση των συνόρων, την ασφάλεια τη αεροπορία και των αεροδρομίων και μιλήσαμε και για το πώ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους Λιβανέζους προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικέ για την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση. Και πρέπει να σα πω ότι τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Όσον αφορά την απειλή τώρα, όπως είπα και αρχικά, πρέπει να μην ξεχνάμε τις παραδοσιακές ε, αδυναμίες ε, των ε, θεσμών στον Λίβανο. Και σε αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνονται και οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, τις οποίες εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Η σταθερότητα της χώρας πάντοτε εξαρτιόταν ε, από ε, άλλους παράγοντες και από τρίτες χώρες. Πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε το, το ζήτημα της διαμάχης μεταξύ Σιητών και Σουνιτών που βρίσκονται, ε, το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών διαμαχών και διαφορών στη Μέση Ανατολή. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε όταν εξετάζουμε τη θέση της Χεσμπολά. Πρόκειται για ένα υπαρξιακό θρησκευτικό ζήτημα. Ε, η μάχη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην, στη Συρία βασίζεται σε αυτά τα υπαρξιακά θέματα. Τα Ισλαμιστικά κινήματα υπάρχουν στην Τρίπολη εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι νέο στοιχείο αυτό. Πρόκειται για ομάδες οι οποίες αποτέλεσαν εύκολο στόχο ε, για να συμμαχήσουν με διάφορα ισλαμιστικά κινήματα, η Σάιντα, το, ο καταβλωρισμός Αναλχάουντα, η ε, βόρεια περιοχή επίσης ε, φιλοξενεί διάφορους πυρήνες και υπάρχουν βεβαίως και εντός της χώρας υποστηρικτές του ISIS και, στο, και, και στα βουνά Καλαμούν. Και υπάρχει και ε, ένας θύλακας ε, ε, του ISIS κοντά στα σύνορα με, τη Συρία. Εμείς είχαμε σκοπό να βοηθήσουμε στην εκπόνηση μιας στρατηγικής η οποία θα είχε ως στόχο τον αφοπλισμό όλων των πολιτοφυλακών εντό ενό έτου, Κάτι τέτοιο βεβαίω δεν έγινε. Η Χεσμπολά έχει διατηρήσει ε, τον ε, εξοπλισμό της. Ε, φυσικά η σύγκρουση στη Συρία έχει αλλάξει τα δεδομένα. Το 2012 η Χεσμπολά ξέρετε ότι άρχισε να συμμετέχει επίσημα στην σύγκρουση στη Συρία και είπε, ε, δήλωσε ότι η ανατροπή του Ασάντ θα ε, ε, έπλητε σοβαρά τον Λίβανο. Αυτό είναι το αφήγημα και έτσι η καταπολέμηση των, του Ισλαμικού κράτους και των τρομοκρατικών ομάδων αποτελεί πλέον σχεδόν αποκλειστική ευθύνη, αποκλειστικό έργο της Χεσμολά. Ένας από τους στόχους βεβαίως είναι να, να προλάβει ε, η Χεσμολά τρομοκρατικές επιθέσεις στα δικά της προπύργια και ε, να ε, διατηρήσει τον, τον, τον έλεγχο ε, εμπορικών διαδρομών συναλλαγών όπλων από το Ιράν προς τη Συρία. Στόχος του, βεβαίως, στόχος της Χεσμπολά είναι να διατηρήσει τα προπήριά της, να καθαρίσει ε, τα όρη Καλαμούν από τους ε, μαχητές του ISIS σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και να ε, μην επιτρέψει την πρόσβαση στα όρη και από τις δύο πλευρές των, των συνόρων. Ως απάντηση έχετε, έχουμε δει βομβιστικές επιθέσεις κατά ΣΥΙΤΟΝ και ε, αρχών ασφαλείας το 2013 και το 2014. Ε, το μεγαλύτερο Η μεγαλύτερη επίθεση έγινε στο Τάνα Φασάλ όπου σκοτώθηκαν 30 στρατιωτικοί. Ε, της, ε, ε, του, Λιβάνου. Παρά τις απώλειες ε, μεταξύ των Σιητών, η Χεσμολά δεν έχει υποχωρήσει και εξακολουθεί να παρέχει ένα είδος σταθερότητας στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τώρα, η επιχειρηματολογία των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι θα πρέπει να ε, πολεμήσουν κατά του ίδιου εχθρού, με, με δυνάμεις ε, που έχουν τον ίδιο εχθρό, ακόμη και αν δεν θα ήταν η πρώτη τους επιλογή. Δεν νομίζω ότι οι, ότι οι δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου δεν ε, μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους. Οπότε υπάρχει και ένα ζήτημα επιχειρησιακό. Βεβαίως, Ποτέ δεν έχει υπάρξει αναφορά επίσημη για συνεργασία. Αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ιδεολογικό επίπεδο υπάρχουν ε, σύνδεσμοι μεταξύ της Χεσμολά και των ενόπλων ε, δυνάμεων. Η Χεσμολά έχει επιδείξει προθυμία να ε, ε, συνεργαστεί με τις αρχές ασφαλείας, ιδίως μετά την ε, τρομοκρατική επίθεση τον Νοέμβριο του 2015. Και η Χεσμπολά ε, δεν πηγαίνει σε μέρη όπου θα μπορούσε να, να πληγεί η εξοπιστία της, όπως στην Τρίπολη, στο Άκα, όπου οι ενόπλες δυνάμεις του Λιβάνου καταφέρουν και ελέγχουν με, με, με σχετικά θετικό τρόπο ε, ικανοποιητικό τρόπο τα πράγματα. Εν συντομία για τη Χεσμολά, ο πόλεμος στην Συρία είναι, έχει έναν υπαρξιακό χαρακτήρα και η ήττα των Σουνιτών Ισλαμιστών είναι για αυτούς ζήτημα ζωής και θανάτου. Και πολλοί από τους υποστηρικτές της Χεσμολά πιστεύουν, ιδεολογικά τουλάχιστον, ότι ε, εκτελούν κάποιο θρησκευτικό καθήκον τους. Αλλά για να επανέλθουμε στο Λίβανο ως, ε, ως σύνολο, συνολικά σαν χώρα, ε, εμείς ε, από την πλευρά μας θέλουμε να έχουμε έναν βασικό εταίρο ε, στη χώρα, τη, χώρα αυτή ως βασικό εταίρο στην περιοχή, γιατί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια οι μόνοι που έχουν ωφεληθεί είναι οι εξτρεμιστές. Το σημαντικό ζήτημα λοιπόν που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο τερματισμός του πολέμου στη Συρία, κάτι που θα ωφελήσει την Ιορδανία, την Τουρκία, το Λίβανο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ένα βηματάκι πίσω και να εξετάσουμε την συνολική πολιτική εικόνα και τα συνολικά πολιτικά ζητήματα που διακυβεύονται στην περιοχή. Thank you very much indeed. Now... Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Τον Εκέλαμ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πραγματογνωμοσύνη και τις συμβουλές σας. Προβληματίζουμε όμως ακόμα για την κατάσταση όπως όλοι μας βέβαια. Ο ρόλος της Χεσμολά και τη στρατιωτικής τη πτέρυγα που βρίσκεται ακόμα στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτή η διένεξη σουνητών Σιητών κυρίως και πώς σας φαίνεται η Χεσπολά σήμερα, τι απόψε έχετε μπορεί να την προσεγγίσουμε χωριστά από το Ιράν από όπου δηλαδή λαμβάνει τον οπλισμό η Χεσπολά και τα χρήματα Δεύτερον, είναι γνωστό ότι η Χεσμολά μπορεί να αποτελέσει μια απειλή για το Ισραήλ με συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή. Συνολικά όμως, είναι μια ρεαλιστική επιλογή αυτή μου θυμίζει την συμμαχία Χίτλερ-Στάλιν. Υπάρχει ένα θέμα ηθικό για μας. Μπορεί το ένα κακό να ιτηθεί με τη βοήθεια του άλλου. Έχει αλλάξει η Χεσμολά. Και ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι. Όπως είπατε, η Χεσβολά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου εδώ και καιρό. Τι γίνεται λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Σφρόντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για αυτή τη θαυμάσια παρουσίαση για την κατάσταση στο Λίβανο. Φαίνεται να το ξεχνάμε αλλά ο Λίβανος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα τώρα με τον πόλεμο στη Συρία το ξεχάσαμε γιατί επισκιάστηκε η κατάσταση κάπως τουλάχιστον δικιά μας στη Σκοπιά την Ευρωπαϊκή από το πρόβλημα των προσφύγων και όταν μιλάμε για το Λίβανο μιλάμε μόνο για τον υψηλό αριθμό προσφύγων που καταβλίζονται στο Λίβανο τεράστιος αριθμός σε σχέση με αυτά που κάνουμε εμείς εδώ. Και ξέρουμε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν όσα πρέπει. Δύο ερωτήσεις έχω εγώ. Ήταν ενδιαφέρον καταρχάς σήμερα να ακούσω ότι υπάρχει στενή συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου με τη Χεσμολά. κάτι το οποίο φαίνεται να σταθεροποιεί την κατάσταση και μάλιστα να πυρορίζει το ριζοσπαστικό χαρακτήρα της Χεσμολά που τόσο συζητήσαμε τα τελευταία 20 χρόνια ιδιαίτερα από τη σκοπιά του νότιου γείτονα του Ισραήλ Αναφέρθηκε από τον κύριο Κιλάμ και θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιο ρόλο διαδραματίζει το Ισραήλ σε όλα αυτά. Γιατί από ό,τι ξέρω το Ισραήλ έχει ξεκάθαρη θέση για την κατάσταση στο Λίβανο. Δεν θα επιτρέψει δηλαδή οτιδήποτε θα το απειλήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε σιωπηλά συμφωνούν με τις εξελίξεις μεταξύ Λιβανικών Όπλων και Χεσπολά. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο του Ισραήλ σε όλη αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Jeffrey Van Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι προλαλήσαντες παρουσίασαν τον περίπλοκο χαρακτήρα της κατάστασης και νομίζω ότι καμιά από αυτές τις τρομακτικές οργανώσεις που περιγράψατε δεν έχει απλή δομή. Παρουσιάζουν πολύπλοκα και πολλαπλά στοιχεία με τακτικούς στρατούς, χρήση τρομοκρατικών μεθόδων. Αποτελούν πολιτικές οργανώσεις. Έχουν και μια θρησκευτική πτυχή επίσης. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά Είτε μιλάμε για το ISIS, είτε μιλάμε για την χέσπολα. Ισχύει το ίδιο. Και αυτό που είπε ο κύριος Κίλαμ υπάρχει κάτι το στρεβλό και το ειρωνικό με όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες αντιμάχονται μεταξύ τους. Βέβαια, να δούμε και το πλαίσιο. Δεν έχουμε κάποια αντικειμενική άποψη για την κατάσταση στο Λίβανο για την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αλλά το κύριο στοιχείο εδώ είναι η ασφάλεια των χωρών μας και οι επιπτώσεις αυτής της ε, συνεχούς τραγωδίας Μέση Ανατολή στην ασφάλεια των χωρών μας. Αυτό είναι το δικό μας το συμφέρον. Βεβαίω μιλάμε για τρομοκρατικές επιθέσεις, μιλάμε για τις επιπτώσεις που έχει όλο αυτό το θέμα στην κρίση των προσφύγων. Οπότε πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαρη στην εστίασή μας στο θέμα αυτό. Τώρα, για το πώς θα επιφέρουμε μεγαλύτερη σταθερότητα, ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε αυτή την περιοχή, ώστε ακριβώς να ωφεληθεί η ασφάλεια το χωρό μας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε ενδιαφέρον την άποψή σας για Λίβανο, Ιράκ, Συρία, για όλη αυτή την περιοχή, πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα σε δέκα χρόνια αυτές τις τρεις χώρες και έξω τον κύριο Γκατράταρ. για το ρόλο επέμβασης ή δράσης της Ένωσης σε αυτές τις περιοχές και το ρόλο της. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν χρήσιμο που θα μπορούσε να κάνει η Ένωση για την αντιμετώπιση τη ε, κατάσταση. Δεν εννοώ βεβαίω συναντήσει, διασκέψει κλπ. Όλε αυτέ τι ανοησίε. και το πρακτικό. Νομίζω ότι η Ένωση όπου είναι πλάκη Παλαιστινική αρχή, αλλά χωρί να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη μόχλευση στην Παλαιστινική αρχή, ώστε να αυτή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να επιταχθεί η ειρήνη, συγγνώμη, πρώτα στην ειρηνευτική διαδικασία, α πούμε. Αλλά ξαναρωτάω, πού μπορεί να βοηθήσει, αν μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γέλα Σεντέρ. Μετά εγώ και μετά θα κλείσω ο κατάλογος. Συγγνώμη έτσι, αλλά έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Η κυρία Γιάλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Περίμενα τα τακτικά μέλη ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Είναι πολύ επίκαιρα και ενημερωμένα στοιχεία. Τρεις ερωτήσεις έχω. Καταρχάς, εντάξει, μ' ακούτε, μ' ακούτε, ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε σχέση με την μελλοντική να την πωλήσει, αν υπάρχει μια τέτοια λύση. Με τι τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς τη διαφορά σε σχέση με τη Χεσμολά. Γιατί είδαμε, ας πούμε, τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νταές, του Άισις, που επέτρεψαν την ανάκαμψη του Συριακού καθεστώτος. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω καλύτερα με ποιο τρόπο η Χεσμολά με τις επιθέσεις της κάτι το οποίο ήταν για μας αρνητικό έτσι έχει μετατρέψει αυτή την στάση μέσω σύγκρουση με το ΙΣΙΣ, μέσω επιθέσεων σε κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση στην Σύρια. Αυτό θα ήθελα να μάθω από του εκπροσώπου. Επίση, οι Δρούζοι, Τζουμπλάτ, Σουφέρ, ποιο είναι ο ρόλο του σε αυτή την κατάσταση που είναι τόσο περίπλοκη στο Λίβανο. Και τέλος, για τους πρόσφυγες. Θα πάμε ως αντιπροσωπεία σε λίγους μήνες. Να μου πείτε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση στους καταβλισμούς των προσφύγων. Κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν, αλλά αυτοί που βρίσκονται στους καταβλισμούς δεν είναι απαραίτητα του ISIS, οπότε θα ήθελα λιγάκι να μας το παρουσιάσετε θα να μας το εξηγήσετε. Ευχαριστώ μετά, αμέσως μετά την δολοφονία του Ραφή Χαρίρη. Ήμουν παρατηρήτρια σε δύο γύρους ε, εκλογών στο Λίβανο και ε, παρατήρησα τότε την αύξηση της επιρροής του Hezbollah. Hezbollah. Ήταν δύσκολη περίοδος. Οπότε η ερώτησή μου και στους δύο μιλητές μας είναι η συμφωνία του ΤΑΙΦ σε τι βαθμό έχει σημασία τώρα, πώς εφαρμόζεται από πολιτική άποψη. Μήπως πρέπει να τροποποιηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σταθεροποιήσουμε περαιτέρω το Λίβανο. ο τελικός μας στόχος είναι να υπάρξει ασφάλεια γενικά και κλειδί είναι η σταθεροποίηση του Λιβάνου. Δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια και σταθερότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης πώς ε, είναι η κατάσταση των μη ε, ριζοσπαραστικοποιημένων ε, σουνητικών κοινοτήτων στο Λίβανο. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ανεχόμεθα το Χεσμπόλα παρά το ότι αυτό σημαίνει ότι διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες ε, εξοπλίζουν και χρηματοδοτούν το Χεσμπόλα και στη Συρία και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά, αλλά, πώς επηρεάζει αυτή η παρουσία ορισμένων ε, φιλιρινικών σουνητικών κοινοτήτων. Βεβαίως μια πλευρά είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Και τίθεται το ερώτημα πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Και πρέπει να διερευνήσουμε και άλλες δυνατότητες και όχι απλώς να εξοπλίζουμε περισσότερο τους ΣΥΙΤΕΣ. Πρώτα ο κύρι, η κυρία Αούν και μετά ο κύριος ε, Γκάτ Ράτσα. Η κυρία Αούν, ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσες αλλά και δύσκολες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ορισμένες και παρακαλώ μετά συμπληρώστε. Εφόσον θέλετε. Πολύ θελήσατε να ενημερωθείτε για το πώς αντιμετωπίζει το Ισραήλ τα θέματα αυτά. Θα έλεγα ότι το Ισραήλ αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που έχει για να αποδυναμώσει το Χεσμπόλα ο Ισραηλινός στρατός μέχρι τώρα θεωρούν ότι απειλούνται πολύ περισσότερο από το Χεσμπόλα παρά από το Ισλαμικό κράτος. Με βάση και την ιστορία της περιοχής και πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, θα έλεγα ότι ε, αυτός ο τρόπος ε, δράσης του Ισραήλ είναι πολύ κακός υπολογισμός, γιατί ανα πάσα στιγμή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα. Το Hezbollah τώρα δεν είναι το Hezbollah του 2000, ούτε της δεκαετίας του 90 ή του 80. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς έχει αλλάξει το Hezbollah. να δούμε πώς δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο και ε, ιδιαίτερα μετά την Ισραηλινή εισβολή του 82 και τι έγινε μετά την ε, κατάληξη της ε, σύραξης αυτής και με τι όρους έγινε αυτό κατά την περίοδο του πρώτου πολέμου του κόλπου και έγινε μια διαπραγμάτευση με τη Συρία. Πάρτε το Λίβανο και βοηθήστε μας για το Ιράκ κτλ. Άρα κάποια στιγμή, με βάση κάποια συγκυρία, παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Και θα προσέξατε ότι η παρουσίασή μου ασχολήθηκε κυρίως με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Άρα οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις μπορεί να έχουν ε, πολύ αρνητικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι εστιάζει υπερβολικά το Ισραήλ ε, στη διαμάχη του με το Χεσμπόλα και δεν έχει μια ευρύτερη προσέγγιση. Και το Ισραήλ, να μην ξεχνάμε, τουλάχιστον η παρούσα κυβέρνηση, έχει επίσης ε, πολλές ιδεολειψίες. Τι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Πολλές από τις ερωτήσεις σας θέτουν το θέμα του ότι δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει έναντι των Παλαιστινιακών Αρχών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και εδώ για τις δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πω κάτι παρόμοιο με αυτό που είπα για το Ισραήλ. Η διαδικασία του Όσλο ξεκίνησε εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόκληση του πώς θα υπάρξει ειρήνη. Και αν δούμε ευρύτερα την εικόνα για τη Μέση Ανατολή και τις διάφορες σειράξεις, δεν πρέπει να χάνουμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε δηλαδή, ότι μία από τις κυριότερες σειράξεις είναι η διένεξη Ισραήλ-Παλαιστινίων. Βεβαίως μπορούν να κάνουν για το θέμα αυτό πολλά, οι χώρες της Ένωσης, η Ένωση. Και δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε σχιζοφρενικοί στο πώς αντιμετωπίζουμε το Χεσμπόλα. Έστω και όχι επίσημα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ρόλο που παίζει το Χεσμπόλα, υποστηρίζει τον ε, στρατό του Λιβάνου και μπορεί να εκτιμάται το έργο των ε, λιβανικών ε, μυστικών υπηρεσιών. Αλλά ό,τι κάνουν, το κάνουν λόγω της συνεργασίας και του συντονισμού των προσπαθειών τους με το Hezbollah. Δεν έχουμε και πολύ σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στα στρατόπεδα σύρων προσφύγων στο Λίβανο. Και βέβαια θα ξέρετε ότι ο Λίβανος έχει πικρή πείρα με τους Παλαιστινιακούς καταβλισμούς. Και τώρα έχει και καταβλισμούς σύρων. και οι Λιβανέζοι δεν κάνουν αρκετά, δεν παρακολουθούν αρκετά τους καταβλισμούς αυτούς για να έχουμε κι εμείς μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει και το αυτό ισχύει και με τους Παλαιστινιακούς καταβλισμούς. Δεν τους ελέγχουν ε, οι δυνάμεις του Λιβάνου. Οι Δρούζοι τώρα. Παρά το ότι ε, παίζει ηγεμονικό ρόλο ο Τζουμπλάτ, οι Δρούζοι δεν είναι μία δύναμη ε, απόλυτα συντεταγμένη και δεν μιλάνε με μια φωνή. Βεβαίως ε, οι θρησκευτικές πεπιθήσεις παίζουν το ρόλο τους, αλλά οι Δρούζοι ξέρετε είναι αρκετά ρεαλιστές. Και όπως σας είπα ορισμένοι νέοι Δρούζοι συμμετέχουν σε διάφορες πολιτοφυλακές ε, τις οποίες κατευθύνει το Χεσμπόλα και μάχονται για να περιορίσουν την δράση του ISIS και άλλων ριζοσπαστικών ομάδων. Τέλος, τέλος. Για τη συμφωνία του ΤΑΙΦ. Το ΤΑΙΦ απεικόνιζε την κατάσταση εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή και τη συνένεση που είχε επιτευχθεί σε εκείνη τη συγκυρία μεταξύ των Λιβανέζων, διάφορων ε, περιφερειακών άλλων δυνάμεων και τις κύριες δυνάμεις Τη διεθνούς σκηνής, τις μεγάλες δυνάμεις. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήταν ε, ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ήταν η καλύτερη που μπορούσε να έχει επιτευχθεί και τη στιγμή δεν ήταν βέβαια η βέλτιστη. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει νέα συμφωνία στο Λίβανο, πρέπει να προσέξουμε ούτω ώστε να μην έχουμε κάτι που να είναι χρήσιμο βράχη πρόθεσμα και ιδιαίτερα αρνητικό σε βάθος χρόνου. Το Χεσμπόλα, όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία, είναι απόρρια τη συμφωνία του Ταΐφ γιατί επέτρεψε στη Συρία να ηγεμονεύσει και η Συρία επέτρεψε στο Χεσμπόλα να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σγκατράτερ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, ακούστηκαν ε, πολύ ενδιαφέρουσες ε, ε, ερωτήσεις. Να σχολιάσω από τη δική μου πλευρά ότι χάσαμε μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Τζον Κέρι πριν από λίγα χρόνια. Πλέον η πολιτική προσοχή έχει προχωρήσει. Σήμερα οι κυβερνήσει ανησυχούν πιο πολύ για την ασφάλεια των πολιτών του για τις τρομοκρατικέ επιθέσει και βεβαίω υπάρχει πάντοτε και το ζήτημα του ΝΤΑΕΣ, το οποίο είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων πολιτικών στο Ιράκ. Πρώτον, του, της διάλυσης του στρατού του Σαντάμ. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τα πράγματα και ιστορικά. Αλλά νομίζω ότι η πολιτική ε, προσοχή πλέον δεν επικεντρώνεται στη διαμάχη Ισραηλινών Παλαιστινίων. Έχουν γίνει τόσο μεγάλες επενδύσεις και σε χρήματα και σε διπλωματικό κεφάλαιο και έχουν καταβληθεί πάρα πολλές προσπάθειες οι οποίες έχουν στεφθεί με αποτυχία. Έχει, έχουμε βγάλει πλέον δηλαδή το, το συμπέρασμα ότι έχουμε μόνο αρνητικές ε, επιλογές μπροστά μας. Φυσικά, αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να καταβάλλονται διπλωματικές προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι μας προσπερνούν τα γεγονότα που σχετίζονται με το Ισλαμικό κράτος. Και αυτό νομίζω ότι είναι η υπαριθμόν ένα απειλή στο μυαλό των πολιτικών μας. Και εμείς πιστεύουμε, για λόγους ασφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το κίνητρό μας ε, για το ποιον θα επιλέξουμε ως εταίρο είναι βεβαίως η ασφάλεια των δικών μας πολιτών. Και ο Λίβανος, όπως και άλλες χώρες περιοχής, κατά μία έννοια αποτελούν μια πρώτη γραμμή άμυνας. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος το να βοηθήσουμε τους Λιβανέζους και άλλους. Και έχετε δίκιο. Τις συνδιασκέψεις και συνομιλίες. Όχι, δεν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό. Έχουμε κάποια εργαλεία στη διάθεσή μας, τα οποία προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά στο Λίβανο υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια απτά αποτελέσματα. Πρώτον είναι η διαχείριση των συνόρων, που είναι πραγματικά σοβαρότατο ζήτημα, όπου προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις τέσσερις διαφορετικές αρχές, υπηρεσίες της χώρας, να βοηθήσουν να αναπτύξουν την ικανότητά τους στα σύνορα. Αυτό φυσικά είναι σημαντικότατο ζήτημα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά την τρομοκρατία. Τους βοηθούμε επίσης με συγκεκριμένο τρόπο όσον αφορά την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συνεργαζόμαστε με θεσμούς της χώρας, με τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να επιτύχουν τις ε, ε, διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές είναι οι δράσεις μας στο Λίβανο. Φυσικά ε, πρέπει να αναφέρω και την ασφάλεια των αεροδρομίων και της αεροπορίας και εκεί υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα όπου και ο Λίβανος μπορεί να ωφεληθεί από την συμμετοχή του στα προγράμματα αυτά. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες αυτές ε, θεματικές ενότητες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Στους καταπληκτισμούς των προσφύγων που έχω επισκεφθεί πολλές φορές ε, νομίζω ότι πολλά από τα προβλήματα αποτελούν και μια, έναν αντικατοπτρισμό των ενδοπαλαιστινιακών ε, προβλημάτων μεταξύ Φατάχ και Χαμάς που αντικατοπτρίζονται και στους καταβλισμούς. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες, ε, διάφοροι δυναμικοί παράγοντες οι οποίοι περιπλέκουν την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να εξετάζουμε τη Μέση Ανατολή ως σύνολο. Θα πρέπει να έχουμε στόχο την ειρήνη, την ευμερία και την ασφάλεια στην Μέση Ανατολή δεν είναι αυτή η εικόνα δυστυχώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι στο μέλλον, αλλά σε κάθε περίπτωση την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση την ενδιαφέρει η σταθερότητα στην, στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και έχουμε στην ε, διάθεσή μας τα, μέτρα, τα μέσα και τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις πρόκλησεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος αλλά δύο λόγια μόνο παρακαλώ, ε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Με ανησυχεί το γεγονός ότι αφήσαμε τις επιθυμίες μας να μας καθοδηγούν. Και υπάρχει εδώ μια απολογητική για την Χεσμολά. Η Χεσμολά ευθύνεται για πάρα πολλά από τα δεινά της ε, που έχουν πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση η οποία έχει ε, κάνει έσχη από τη δεκαετία του 80. Την δολοφονία του Ράφη το 2012, την, ε, το, τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στη Βουλγαρία δεν έχουν περάσει και τόσα πολλά χρόνια από τότε που η Χεσμπολά έβαλε ε, έβαψε τα χέρια της με αίμα. Ε, δεν, είναι, πρόκειται, δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια ε, οργάνωση με θετικές προθέσεις, αλλά πρόκειται στην ουσία για το όπλο του Ασάντ και των Ιρανών στο κεφάλι της κυβέρνησης του Λιβάνου. Συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, ο χρόνος μας τελείωσε, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να καταφέρουμε να ξαναζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί είναι ανάγκη να εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τα ζητήματα που απασχολούν το Λίβανο, γιατί εγκαταλείψαμε τη χώρα δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια και δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή. Σας υπόσχομαι ότι θα το βελτιώσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ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 permission. They need to go at 11 o'clock sharp to the airport. Uh-huh. Ladies and gentlemen, please be seated. We have to start immediately. Κυρίες ε, και κύριοι, καθίστε παρακαλώ, πρέπει ξεκινήσουμε αμέσως. Δύσκολα ξεκίνησε η μέρα σήμερα λόγω καθυστέρησης που οφείλεται στο κυκλοφοριακό, οπότε χρειάστηκε να επιταχύνουμε. Να ξεκινήσουμε αμέσως λοιπόν με το επόμενο σημείο της ημερησιάς μας. που αφορά ένα από τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η υποεπιτροπή μας. Δηλαδή, αξιολόγηση και αποτίμηση του ρόλου των Αποστολών της Ένωσης όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας στην Ουκρανία με την EU AM τη συμβουλευτική δηλαδή αποστολή της ΕΕ και εκεί θα αξιολογήσουμε λοιπόν την δράση της EUAM και τις προοπτικές όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις εκεί στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας μεταρρυθμίσει που γίνονται με τη βοήθεια της ΕΕ και το ρόλο της EUAM. Χαίρομαι λοιπόν που καλωσορίζω έναν θαμώνα εδώ της υποεπιτροπής μας, τον Kenneth Dean, διευθυντή του CPCC από την ΑΕΔ, σχεδιασμός και διεξαγωγής δηλαδή επιχειρήσεων Έχουμε και την επικεφαλή τη αποστολή τη EUM στην Ουκρανία και στου τη Λαντσίσκα. Αποστολή που πήγε στην αρχή του χρόνου στο Κίεβο φέτο. Με χαρά λοιπόν σας καλωσορίζω. Και τέλος, τον επικεφαλή της Γιώργη Γέλιν, μάλλον καλωσορίζω, πρεσβευτής της Ουκρανίας. Ο κύριος Τουτσίνσκι δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Ο επικεφαλής αντιπροσωπείας δηλαδή της Ουκρανίας στην ΕΕ. Και καλωσορίζω ανταυτού τον κύριο Γέλιν. Εδώ. Στο βήμα. Να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Γέλιν για μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης στην Ουκρανία που αφορά την ασφάλεια. Μετά ο Κενεθ Ντίν θα μας μιλήσει για σημαντικά επίσης ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια. Και μετά θα έχουμε μια πλήρη και διεξοδική παρουσίαση των δράσεων της EUM στην Ουκρανία από την κυρία Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ στην εκδήλωση αυτή. Όπως ξέρετε, εδώ η κατάσταση στην Ουκρανία είναι κάπως υβριδική. Ο στόχος, όπως και ο Πάπας, δεν είναι ένας τρεις παγκόσμιος, αλλά ένας τρεις παγκόσμιος και καλυμμένος. Δηλαδή, έχουμε τις ΗΠΑ οι οποίες προσπαθούν να να προσελκύσουν την Ευρώπη και να δράσουν στην Ουκρανία. Το πιο ευαίσθητο θέμα εδώ είναι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να ασχοληθούμε με τον επιδιθόμενο και να αντιμετωπίσουμε τις μεταρρυθμίσεις ταυτόχρονα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ως έθνος πώς θα επιβιώσουμε. Βασιζόμαστε λοιπόν στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς είχαμε τις κυρώσεις προς τον επιτιθέμενο. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την παραβίαση εθνών κανόνων και Ξέρω ότι υποφέρουν οι εταίροι μας από τα αντίμετρα των Ρώσων, αλλά πιστέψτε με, αν η Ρωσία καταφέρει να κατακτήσει την Ουκρανία, θα πρέπει να πληρώσετε τα εκατονταπλάσια. Και η ασφάλεια προέχει. Έχουμε κάποια κριτήρια τώρα για εκλογές που θα διασφαλίζουν ε, την ε, ασφάλεια μετά το Μάρτι Τώρα για την κατάσταση ασφάλειας επιτόπου στη χώρα μας. Θα πρέπει να το δείτε κατηδίαν. Έχουμε και την εμπλοκή του ΟΗΕ. Και να σας πω και τα εξής. Στόχο μας για φέτος είναι το να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των θεσμών μας. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν την αδιαφάνεια, τη διαφθορά, κάνουμε ελέγχους ακεραιότητας και θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα γενικό γραφείο επιθεωρητή που θα λαμβάνει υπόψη του την εμπειρία των ΙΠΑ σε αυτό το τομέα. Αυτό θα δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Είχα πάει στην Περσιόνα στην Ιταλία πριν μια εβδομάδα. Κοιτάζουμε και άλλα ενδεχόμενα, όπως ε, διαμεσολαβητής, ε, συνεργασία στενή τα κτλ. Μετά, διακυβέρνηση, πιο το οχι. Θέσπιση επίσης κριτηρίων για την επιλογή των εισαγγελέων και των δικαστικών. Οι αρμοδιότητές τους, όλα αυτά θα μεταβαστούν ως δικαιοδοσίες στα ερευνητικά σώματα. Επίσης να πω ότι πρόσφατα συνάντησα τον κύριο την κυρία Λαντσίσκας και συζητήσαμε σύντομα και είπαμε ότι οι προτεραιότητε μας είναι κοινέ και τι επόμενε εβδομάδες επίσης θα καταρτήσουμε ένα κατάλογο δράσεων για τον οποίο βέβαια θα σας ενημερώσω όσον αφορά τι υψηλέ προτεραιότητε. Θα έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης και βεβαίω βασιζόμαστε στη δικιά σα την εμπειρία και πραγματομοσύνη. Πριν δύο εβδομάδες ε, περάσαμε και ένα νόμο για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης τεράστιας σημασίας, οπότε βασιζόμαστε στην εμπειρία σας. Επίσης, θα θέλαμε να βελθούμε και από την δικιά σας την εμπειρία όσον αφορά την παρουσία εισαγγελέων και άλλων δικαστικών λειτουργών στην περιοχή. Εγώ πάντως θα, θα προσπαθήσω να σας παράσχω τις ε, καλύτερες πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου και νομίζω ότι πολλά θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού. Πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο της ε, παρουσίας της Αποστολής της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελέα για την πολύ σύντομη και περιεκτική παρουσίαση. Ο κύριος Κένεθ Ντίντορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που στείλατε για να μιλήσουμε για την ε, πολιτική αποστολή στην ε, Ουκρανία. Η Ουκρανία παραμένει πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από πλευρά ασφαλείας, αλλά και ευρύτερα πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και χαιρόμεθα που μπορούμε να βοηθήσουμε να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις. Θα ασχοληθώ με δύο-τρία βασικά σημεία πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που θα σα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε τον προηγούμενο Ιανουάριο σας είχα μιλήσει στο μέλλοντα χρόνο για το τι θα μπορούσε να κάνει η αποστολή μας για να συμπληρώσει την στρατηγική κεντρική εντολή που είχαμε έκτοτε ο κύριο Λαντσίσκας που έχει οριστεί το Φεβρουάριο χαίρομαι που μπορώ να σας τον παρουσιάσω σήμερα ήταν επικεφαλής αποστολή στο Βίλνιους έχει πολύ πείρα ως ε, αστυνομικός και πολύ πείρα προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και αυτά που έχει κάνει σχετίζονται με αυτά που θέλουμε να κάνουμε στην Ουκρανία. Χαιρόμεθα πολύ που έχουμε λοιπόν ένα τόσο έμπειρο και υψηλού επίπεδου υπεύθυνο για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις σοβαρές προκλήσεις. Ποια είναι η εντολή. Συμπληρώνει αυτά που κάναμε προηγουμένως σε κεντρικό επίπεδο, με συγκεκριμένα στοιχεία, βήματα. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι μας ζήτησαν τα κράτη-μέλη. Μας ζητούν ακόμη να συμπληρώσουμε την στρατηγική ε, κεντρική ε, βοήθεια που δίνουμε, να βοηθήσουμε τη δημόσια την αστυνόμευση, την τοπική αστυνομία, καλύτερη, καλύτερο συντονισμό χωρίς αρμοδιοτήτων, καλύτερες εσωτερικές δομές και με, ε, και με την αστυνομία, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, να βοηθούμε περισσότερο στις ποινικέ έρευνες, όπως ανέφερε και ο Σαγγελέας. Ο, ο συνάδελφος μου θα σας πει περισσότερα για όλα αυτά. Όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν την επαφή μεταξύ του πληθυσμού με τους αστυνομικούς και η τοπική αστυνομία δεν έχει εύκολο έργο. Έχει έργο να ασχοληθεί με διάφορα χωριά, μικρές πόλεις. Η τοπική αστυνομία, ο κύριος στόχος της είναι να μπορεί να έχει στενή επαφή, να μιλάει με τον πληθυσμό μια αποτελεσματική αστυνομία πρέπει να έχει αποδοχή από τους αστυνομευόμενους και να εργάζεται σε συνεργασία με αυτούς. Αυτή η αποδοχή είναι βασική για οποιαδήποτε αστυνομία που θέλει να παράσχει σωστές υπηρεσίες. Για να αποτελεσματική η αστυνόμευση είναι πιο σημαντική από την ίδια την αστυνομία. Η αστυνόμευση σημαίνει οι κάτοικοι να βοηθούν τους αστυνόμους να διατηρούν την τάξη, να προτρέπουν ε, να μην γίνονται παράνομες πράξεις. Γι' αυτό θέλουμε να συνεργαζόμεθα με την εισαγγελία. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει αυτή η συνεχή σχέση από το πρώτο σημείο επαφής του αστυνομικού με έναν κάτοικο μέχρι όλη τη δικαστική διαδικασία, είτε είναι θύμα, είτε είναι ε, μάρτυρας, να αντιμετωπίζεται σωστά, να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να μην του αρνούνται την πρόσβαση, ακόμη και αν είναι ε, κατηγορούμενος. Ελπίζει η Ένωση, αναμένει η Ένωση ότι η Ουκρανία θα το επιτύχει αυτό. Βεβαίω είναι δύσκολο. Πρέπει να δημιουργήσουμε την εμπιστοσύνη των κατοίκων ε, στις υπηρεσίες ασφαλείας και η αστυνομία της Ουκρανίας πρέπει να προστατεύει τον πληθυσμό. Δεν πρέπει να είναι λοιπόν επιθετική, δεν πρέπει να τρομοκρατεί τον πληθυσμό. Πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των κατοίκων. Και αυτό δεν γίνεται εύκολα. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες. Πρέπει να αλλάξει αντιμετώπιση. Χρειάζεται να υπάρχει ισχυρή ηγεσία από το Υπουργείο μέχρι τον επικεφαλής κάθε αστυνομικού τμήματος θα τα πει ο συναδελφός μου, έχουν κάποια προγράμματα συγκεκριμένα στο Χάρκιβ και αλλού, όχι μόνο στο Κίεβο λοιπόν, ε, δουλεύουμε σε διάφορες περιοχές. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, κύριε Ντίν. Βλέπω ότι είναι μαζί μας ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, ο κύριος Βιτάλη Λουτσέγκο και γνωρίζω ότι δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του γιατί πρέπει να προλάβει την πτήση του. Ε, ελπίζω να προλάβω να του δώσω το λόγο για ένα λεπτό μετά τον κύριο Λαντσίνσκας. Θα συνεχίσω στα πολωνικά και θα... Όχι μάλλον. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο στον επικεφαλής της EUAM, τον κύριο Λανσίνσκα. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Πολύ σύντομα θα παρουσιάσω σε εσά ε, την αποστολή μας στην Ουκρανία. Η αποστολή μας δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Ε, είναι μια αποστολή μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Οι δραστηριότητε της αφορούν την στρατηγική συμβουλευτική, την ε, βοήθεια στον ε, τομέα της ασφάλειας όσον αφορά την ε, υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η τρίτη είναι ο συντονισμός και η συνεργασία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε πέντε προτεραιότητες, τις οποίες έθεσαν τα κράτη-μέλη, πέντε γραμμές δηλαδή. Πρώτον είναι η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, δεύτερη είναι η αστυνόμευση, τρίτη η δημόσια τάξη, οι ποινικέ έρευνες είναι η τέταρτη και η πέμπτη είναι η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Και φυσικά έχουμε τρία οριζόντια ε, θέματα που μας απασχολούν, καλή διακυβέρνηση, καταπολέμηση διαφθοράς και ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα φύλου. Τι κάνουμε τώρα. Από τις 11 Μαΐου ε, ε, έχουμε παρουσία σε τρεις περιοχές, η έδρα μας είναι στο Κίεβο και έχουμε δύο περιφερειακά γραφεία στο Χάρκιβ και στο Λιβύβ. 17 υπαλλήλου έχει η αποστολή μας σε κάθε γραφείο. Τι κάνουμε. Παρέχουμε εκπαίδευση σε αστυνομικές σχολές, και παρέχουμε συμβουλές για το πώς μπορούν να καταστούν οι αρχές αποτελεσματικότερες και να διαχειρίζονται τους πόρους τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε και κινητές μονάδες, οι οποίες ε, επεμβαίνουν σε ad hoc βάση και έχουν συμμετάσχει σε κάποια ε, εκπαιδευτικά σεμινάρια μικρής κλίμακης ε, σε περιοχές όπου δεν έχουμε μόνιμη παρουσία. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Έχουμε συνεργασία με την Εθνική Αστυνομία. Έχουμε συστήσει τέσσερις ομάδες εργασίας για διάφορους τομείς, για την, την, τον επανεξέταση των αστυνομικών, ε, για ζητήματα χρηματοδότησης, καλής διαχείρισης, χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, ε, προγράμματα αστυνόμευσης ε, και ε, βοήθεια προς, τις, προς την Εθνική Αστυνομία της χώρας για την διαχείριση μεγάλων όγκων ανθρώπων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις ανοιχτές. Ναι, κύριε Εισαγγελέα, δυστυχώς πρέπει να φύγετε, το γνωρίζω. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά που βρεθήκατε εδώ μαζί μας. Yes, please, please just... Oh. Thank you very much. Ευχαριστώ. Όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ε, μεταρρύθμιση στην Ουκρανία. Ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά μου, διότι ως πολιτικός κρατούμενος ε, τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερα να τα εξασκήσω. Αυτό που ε, ενδιαφέρει εμάς είναι η αλλαγή των, καθηκόντων του Γενικού Εισαγγελέα. Έχω δύο βασικά καθήκοντα πλέον. Να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη του Ουκρανικού λαού, το οποίο θα επιτευχθεί μέσω της καταπολέμησης διαφθοράς, της εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος και της δίωξης όσων κατέστρεψαν την εμπιστοσύνη του ε, ε, ουκρανικού λαού. Και τέλος και δεύτερον να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα διαφθοράς. Στην Ουκρανία δεν έχουμε διαφθορά, αλλά έχουμε οργανωμένο έγκλημα. Κάθε αλλαγή πολιτικής φρουράς πριν την Επανάσταση αλλά και μετά την Επανάσταση δεν άλλαξε ποτέ αυτό το όνειδος του οργανωμένου εγκλήματος. Εμάς δηλαδή μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ψάρι, αυτό το, το μεγάλο πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος. Και ελπίζω στο τέλος της φετινής χρονιάς να ξαναβρεθούμε και να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε θετικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι είναι το τελευταίο κύμα αυτό που βιώνουμε τώρα ε, του πολιτικού συστήματος μετά την επανάσταση του Μαϊντάν. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους, ε, α, α, τους, ε, τους ομιλητές και ιδίως αυτούς που ανέφεραν ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας δεν έχει την απαραίτητη κατάρτιση στόχος του εισαγγελέα είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Ναι, εγώ δεσμεύομαι ότι θα απαλλάξω το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας από κάθε πολιτική επιρροή. Είναι στόχος μου, είναι το καθήκον μου, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή μου ώστε σε συνεργασία με τους δυτικούς φίλους μας, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαγγελέα για αυτήν την πολύ ειλικρινή δήλωσή σας. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ξέρω ότι έχουν ζητήσει ήδη κάποια μέλη το λόγο. Θα μιλήσουν ο κύριος Λουτσίσκας, ο κ. Κένευθυντίν. Το βασικό ζήτημα που αφορά την, τις αρχές ε, επιβολής του νόμου είναι η ωρεοθέτηση των αρμοδιοτήτων. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία έχουν προχωρήσει και χάρη στην αποστολή EUAM με τον τωρινό αλλά και τον προηγούμενο επικεφαλής της. Βεβαίως θα θέλαμε οι μεταρρυθμίσεις αυτές να επιταχυνθούν, αλλά συμμερίζουμε αυτό που είπαν οι Ουκρανοί συνάδελφοι, ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση μια χώρα να διαφυλάσει την εδαφική της εκαιρεότητα και ταυτόχρονα να διέρχεται από τόσο δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Με πρακτικούς όρους, ποιο είναι το, όριο, το, το όραμα της οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων. Ποιες είναι οι συμβουλές που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομέα. Ποιες αρμοδιότητες θα πρέπει να κατανεμηθούν σε ποια κρατική αρχή. Και πώς θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία και τη σύσταση αυτών των ε, αρχών ε, και υπηρεσιών. Ο λόγος ε, στην κυρία Λόζιν. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας. Ναι, είναι πράγματι ε, πάρα πολλά τα πράγματα και πολύ περίπλοκα. Αναφέρθηκαν τα, τα ζητήματα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, οι μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ε, εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση των αρχών επιβολής του νόμου. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω την έκθεση του ΥΠΑ του ε, αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ το 2015 έγιναν 1.900 καταγγελίες ε, στη Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας για βασανιστήρια από αστυνομικού. Αλλά μόνο σε 49 από αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε καταδίκη. Αυτός ο υψηλός αριθμός δεν δείχνει τουλάχιστον ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία της Ουκρανίας συνεχίστηκε τουλάχιστον ε, μέχρι και το 2015 σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μιας και έχουμε εκπροσώπους της χώρας εδώ, πώς εξηγείτε εσείς τον πολύ μικρό αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων. Ποια είναι η δική σας γνώμη και ποια είναι η γνώμη της EUAM για αυτό το θέμα και ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε από τα στοιχεία αυτά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Αντρική Ένα, από το ΕΛΚ. Δεν είχα δει το έτοιμά σας για το λόγο. Συγχαρητήρια κιόλα. Νέο μέλος που αντικαθιστά από ό,τι θυμάμαι τον κύριο Λανσπέρκης. Έχετε το λόγο. Και μετά κυρία Χάμψα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. χαιρετίζω τον κύριο Λαντσίσκα και τον κύριο Λουτσένκο, τον εισαγγελέα συμπατριώτες. Να αναφερθώ στα κύρια προβλήματα της Ουκρανίας, όχι μόνο δηλαδή η διαφθορά, αλλά το σύστημα εγκληματικότητα που φτάνει στα υψηλότερα κλιμάκια της χώρας Μιλήσατε για την ανεξαρτησία του Γενικού Συγγελέα. Πώς θα το πετύχετε. Βεβαίως, εμείς καλωσορίζουμε αυτή την πρόθεση, όπως και ο λαός, αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Τι θα κάνετε για να το πετύχετε. Ευχαριστώ κύριε Χάρμς. Ε, ε, λοιπόν, ακούστε με και εμένα στα γερμανικά. Ευχαριστώ τους ε, κυρίους από την Ουκρανία και θέλω να τους συγχαρώ για αυτά τα οποία έγιναν για την ε, διατήρηση της ειρήνης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την περασμένη Κυριακή στην Ουκρανία, στο Κίεβο συγκεκριμένα. Ήταν αυτή η διαδήλωση για την οποία υπήρξε πολύ σωστή προστασία των ε, συμμετεχόντων. Ήταν η πρώτη ε, διαδήλωση Gay Pride στο Κίεβο και υπήρχε πολύ σωστή παρουσία της αστυνομίας, ε, πολυάριθμη, για να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμμετεχόντων. Όλοι όσοι συμμετείχαμε από την Αντιπροσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντυπωσιαστήκαμε από αυτά που είδαμε την περασμένη Κυριακή στο Κίεβο. Είδαμε ότι η παρουσία της αστυνομίας, που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν υπερβολική, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σύμβολο αυτό, ότι η αστυνομία είναι διατεθειμένη να παίξει το ρόλο της ε, και τον ε, βλέπει τώρα διαφορετικά το ρόλο της. Είναι λοιπόν μια σαφής απτή εκδήλωση ότι αλλάζουν τα πράγματα. Οι ερωτήσεις προκύπτουν από τον τίτλο της συζήτησης. Ε. Θα ήθελα να μου πείτε εάν η οξυμένη κατάσταση ασφαλείας ε, ε, στα ανατολικά της χώρας που έχει προκύψει από την αύξηση των επιθέσεων των ε, αποσχιστών θα έχει επιπτώσεις στις προσπάθειες μεταρρύθμισης των δυνάμεων ασφαλείας. Γιατί, όχι αδίκως, συχνά αναφέρεται, ότι η Ουκρανία πρέπει να εισαγάγει αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση είναι μια χώρα που δεν αποφάσισε να επιβάλλει κατάσταση πολέμου. Είναι μια χώρα που πρέπει να αφιερώσει πολλέ δυνάμει ασφαλεία και αστυνομία και στρατό στην προσπάθεια καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Ρωτάω λοιπόν, η οξυμένη κατάσταση κατά μήκο τη λεγόμενη αποστατικοποιημένη ε, ζώνη, ρωτάω λοιπόν αν έχει επιπτώσει στι προσπάθειε μεταρρυθμίσεων το Σαββατοκύριακο ήμουν εκεί και μίλησα και με την ε, ε την ε, διαμεσολαβήτρια για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Ουκρανικές αρχές. Οπότε, θα ήθελα να μάθω τι προσπάθειες έχουν γίνει για να γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις διότι το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Ουκρανία η Επιτροπή που ήταν εκεί για την παρακολούθηση των ε, βασανιστήριων είναι κακό μήνυμα. Ο κύριος Οστρεβίτσιος, ε, πρόεδρος των φίλων της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους και καλωσορίζω τους αξιωματούχους και φίλους από την Ουκρανία. Εμείς πραγματικά εκτιμούμε αυτά τα αποφασιστικά βήματα προς μεταρρύθμιση των συστημάτων ασφάλειας και δημοσίων αρχών. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση που κληρονομήσατε μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Είχα μια κατάσταση αστάθειας και την παρουσία πρακτόρων από την ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Ακούσαμε να γίνεται εκτενός λόγος γι' αυτός. Δεν είχαμε μόνο την διείσδυση της αντικατασκοπίας, αλλά και την παρουσία σε δημόσιες αρχές, στα Υπουργεία και αλλού. Κινούσαν τα νήματα από το παρασκήνιο και γι' αυτό θέλω να θέσω το πρώτο ερώτημα κατά πόσο τα συστήματα ασφαλείας της Ουκρανίας προστατεύονται ή έχουν ε, γίνει πια στεγανά σε σχέση με τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Ένα άλλο θέμα που συζητάμε είναι το εξής. Πηγαίνουμε σε ένα καθεστώς ελευθερία στην Ουκρανία και υπάρχει ένας μηχανισμός και ένα νέο κανονισμός που προετοιμάζεται ώστε να επιτηρείται η κατάσταση που αφορά το εαυτό ελεύθερων θεωρήσεων για την Ουκρανία. Βεβαίω ακούσαμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, διαφθορά κτλ. Εγώ είδα κάποιε θετικέ στατιστικέ και μια και εξέφρασαν ανησυχία οι Γερμανοί συνάδελφοι ότι κάποιοι υπήκοοι κάποιων χωρών ε, συνεισφέρουν στην εγκληματικότητα. Από το 2015 οι εκθέσει της Ρημανικής Αστυνομίας θέτουν τους Ουκρανούς στην 23η θέση όσον αφορά την εγκληματικότητα. Ερωτώ λοιπόν, κατά πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει την σημασία της προετοιμασίας για αυτή την απελευθέρωση ή φιλελευθερωποίηση και τι γίνεται με τα γραφεία της αστυνομία, του εισαγγελέα και άλλων αρχών που βρίσκονται υπό έρευνα ώστε ακριβώς να εφαρμοστεί σωστά το καθεστώς ελεύθερης θεώρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτρας. Να προσθέσω μόνο ότι εξίσου και η Γεωργία βρίσκεται χαμηλά σε αυτό τον κατάλογο που ανέφερες παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω τους εξέχοντες Ουκρανούς εκπροσώπους στην συνάντησή μας. Μια σύντομη παρατήρηση έχω μόνο. Να ευχαριστήσω την Ουκρανία για αυτό που έχει κάνει ώστε να προστατεύσει την Ευρώπη από την τρομοκρατία. με τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι μυστικές αρχές των, της Ουκρανίας για τεράστιες ποσότητες οπλισμού. Αυτό που κάνατε αποδεικνύει ότι η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας έχει νόημα όσον αφορά την ασφάλεια και την αντιμετωπίση της θερμοκρατίας σε μια περιοχή όπου είμαστε σχετικά ευάλωτοι μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ και πάλι και να πω ότι σας επικροτώ επειδή συζητήσαμε για τις λεπτομέρειες αλλά όταν ένας εταίρος μας ε, συλλαμβάνει τρομοκράτες με τέτοια ποσότητα οπλισμού και μετά προσφέρει αυτές τις πληροφορίες στην Ένωση η Ένωση δεν μπορεί παρά να ευχαριστήσει τους εταίρους της που το έκαναν αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρη. Τώρα να ζητήσω από τους ε, ομιλητές μας να απαντήσουν στα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις. Λαντσίσκας πρώτα και ο Κύριος Λουτσάνη και ο κ. Ντίν. Βεβαίω, αν θέλει να λάβει και το λόγο, ευχαρίστω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα και μετά θα δώσω το λόγο στο Γενικό Εισαγγελέα για να απαντήσει για ερωτήσει που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένε ε, δικαστικέ έρευνε, όπω είπα η αποστολή μα, είναι μη εκτελεστική. Χορηγούμε πολύ κατάρτιση στους αστυνομικού, στους υπαλλήλου των εισαγγελιών, όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και στην επαρχία. Και κυρίω ασχολούμεθα με την τοπική αστυνόμευση. Με την ευρύτερη έννοια προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, θέματα ισότητας φύλων, όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά και των ε, παθών, των θυμάτων, όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση. Ξέρετε, είμαστε σε μεταβετική περίοδο και ορισμένες φορές ε, συμβαίνουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν παραπτώματα, αλλά κάνουμε πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και πραγματικά την παρακολουθούμε. Το καλό παράδειγμα ήταν αυτή η εκδήλωση την Κυριακή, αυτή η εκδήλωση για την ισότητα όπου η αστυνομία έλαβε υπόψη τις συμβουλές μας και έδρασε, ανέλαβε πρωτοβουλίες και ήταν πραγματικά μεγάλη επιτυχία η αστυνομική πλαισίωση αυτής της εκδήλωσης. Για τα θέματα τώρα αρμοδιοτήτων έχουμε την Εθνική Αστυνομία, που κάνει 90% των ερευνών <clears throat> και ανακρίσεων, <clears throat> οι υπηρεσίες κρατικής ασφαλείας που είναι αρμόδιες για ορισμένες ε, έρευνες, έχουμε την υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς και την ε, νέα υπηρεσία <clears throat> ερευνών που θα αρχίσει να λειτουργεί μέχρι τέλος του χρόνου. Και άρα υπάρχει θέμα οριοθέτησης αρμοδιοτήτων που είναι δική μας αρμοδιότητα, η εισαγγελία. Η εισαγγελία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό όλων των ποινικών ανακρίσεων και ερευνών. Για το SSU που είναι οι υπηρεσίες κρατικής ασφαλείας συνεργαζόμαστε με τους ε, Ουκρανούς εταίρους μας για να υπάρξει μεταρρύθμιση των ε, υπηρεσιών ασφαλείας. Αλλά ξέρετε, τέτοιου είδους υπηρεσίες ε, δεν είναι εύκολο να μεταρρυθμιστούν. Ήδη λειτουργούν πλήρως και έχουν λόγω της πολιτικής κατάστασης πολλή δουλειά. Και πρέπει επίσης να κάνουν και μεταρρυθμίσεις και αναδιοργάνωση και να υπάρχει και έλεγχος, δημόσιος έλεγχος. Και επίσης, όπως σας είπα, κάνουμε πολύ κατάρτιση, εκπαίδευση. Ε, έρχονται οι υπάλληλοι από την Ουκρανία και οι αστυνομικοί στο Europol. Τους ενημερώνουμε για θέματα προστασίας στοιχείων, γιατί είναι πολύ βασικό να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά με ασφαλή τρόπο βέβαια. Και έχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λουτσάνκα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε. κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, συμβαίνουν, ναι. Η υπηρεσία μου έχει λάβει ένα περιοδικό από τις φυλακές. Α, όχι, συγγνώμη, είναι ίσως ένα φλιτζάνι από τις φυλακές. Το φλιτζάνι που είχα εγώ, έχω η υπηρεσία μου, το έχω δώσει στην υπηρεσία μου, το φλιτζάνι που είχα εγώ όταν ήμουν πολιτικός κρατούμενος. Και για να θυμόμαστε ότι έχουμε ακόμη πολλούς που είναι προφυλακισμένοι χωρίς να έχουν ε, ε, ακόμη ημερομηνία για τη δίκη τους και που έχουν προβλήματα υγείας. Έχω ένα κατάλογο από την κυρία ε, λαβήτρια για ορισμένους οι οποίοι περιμένουν 4, 10, 12 χρόνια. Αλλά αυτοί θα απελευθερωθούν τώρα. Θα αλλάξουμε τον ανώτατο χρόνο προφυλάκησης. Και ορισμένοι που έχουν σοβαρά προβλήματα, για παράδειγμα ε, με σοβαρά προβλήματα καρδιακά και τέτοια, όπως έγινε και με μένα και τη Γιούλια Τιμοσέγκα παλιότερα. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο η καταπολέμηση τη εγκληματικότητα, αλλά και η τήρηση, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί έχω προσωπική πείρα. Ναι, οι συνθήκε κράτηση είναι πολύ κακέ. Εγώ και η Γιούλια Τιμοσέγκα Είμαστε κρατούμενοι σε φυλακές ε, του 19ου αιώνα. Ήταν άθλια η κατάσταση. Αλλά χρειαζόμαστε, ξέρετε, πόρους ε, για να επισκευάσουμε τις φυλακές. Αλλά δεσμεύομαι προσωπικά. Θα αλλάξω τις συνθήκες κράτησης, όπου χρειάζεται. Έχω διορίσει έναν ε, νέο αρμόδιο στη Γενική Εισαγγελία για τις φυλακές και επίσης ε, προηγουμένως ήταν στην υπηρεσία της διαμεσολαβήτριας και τώρα είναι υπεύθυνος για τις φυλακές. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα ε, καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Να σας δώσω παραδείγματα. Βεβαίω έχουμε μια χωριστή υπηρεσία για την αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ε, υπηρεσία για την καταπολέμηση διαφθοράς. Και αυτό το μήνα δημιουργήσαμε ένα νέο Ουκρανικό Γραφείο Ερευνών. Όλες τις έρευνες θα τις κάνει αυτή η νέα υπηρεσία όλες τις νέες υποθέσεις. Αλλά τις παλιές υποθέσεις για τα επόμενα δύο χρόνια θα την έχει το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας. Και κατόπιν θα σταματήσει η Γενική Εισαγγελία να κάνει έρευνε. Αλλά για αυτά τα δύο χρόνια θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος όπου συμμετέχουν και ανώτατοι υπάλληλοι. Δεν είναι μόνο θέμα του Γιάννου Κόβιτς, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ο Γιαννουκόβιτς έχει κλέψει δις, δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα κάθεται στη Μόσχα. Αλλά δεν τα έκανε μόνος του. Το δίκτυό του οργανωμένου εγκλήματος είναι ακόμη στην Ουκρανία και ορισμένοι από αυτούς συμμετέχουν να κλέβουν στην εφορία, στα τελωνία. Οι φυπουργοί είναι ορισμένοι, ανώτατοι αστυνομικοί, εισαγγελείς και κλπ. Άρα η καταπολέμηση της μαφίας του Γιαννουκόβιτς πρέπει να συνεχιστεί. Ένα μικρό παράδειγμα. Θεωρούμε ότι έχουν κλέψει από την επιχείρηση φυσικού αερίου 700 εκατομμύρια ευρώ. Την προηγούμενη εβδομάδα Δέκα μέρες μετά την ανάληψη αρμοδιοτήτων από πλευρά μου έγιναν δύο συλλήψει. που θεωρούμε ότι είναι υπεύθυνοι για αυτήν την υπεξαίρεση από τον κρατικό προπολογισμό. Νομίζουμε ότι έχουν δύο εργοστάσια τσιγάρων και επίσης μια λυσίδα βενζινάδικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έχουμε στοιχεία, θα σας τα παράσχουμε και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε πίσω αυτά τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Και δεν κάνουμε διακρίση μεταξύ των παλαιών εγκληματιών και των νέων, γιατί δρούν ε, μέσω του ιδίου συστήματος. Βεβαίως έχω μακρά πείρα ως πολιτικός. Ίσως να έχω ένα πολιτικό βάρος στη χώρα μου. Θα αξιοποιήσω λοιπόν κάθε δυνατότητα που έχω ούτως ώστε η εισαγγελία να είναι ανεξάρτητη και διατεθειμένη να στραφεί κατά οποιοδήποτε πολιτικού, οποιοδήποτε υπευθύνου από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας που να ανοίξει οποιοδήποτε κόμμα και που θα εργάζεται σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Τρίτον, εάν τα συστήματα ασφαλεία μας ε, προστατεύονται από την προσπάθεια των Ρώσων να διεισδύσουν. Τώρα καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί θυμάμαι ότι παλιά ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας μας ήταν Ρώσος πολίτης. Ο Υπουργός Χάμινας ήταν Ρώσος πολίτης. Και άλλοι. Ο επικεφαλής των σωματοφυλάκων του Προέδρου Γιαννουκόβιτς ήταν Ρώσος πολίτης. Τώρα λοιπόν υπάρχει περισσότερη προστασία. Αλλά δεν έχει τελειώσει αυτή η προσπάθεια. Απελευθέρωση θεωρήσεων. Μπορώ να σε εγγυηθώ ότι τα στοιχεία που θα σας στέλνουμε, τα έγγραφα που θα σας στέλνουμε θα είναι προστατευμένα. Απόλυτα ασφαλή. Καταπολέμηση γενικότερα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, δεν θέλω να πω περισσότερα. Γιατί το ζήτημα είναι ε, να δράσω και όχι να κάνω διακηρύξεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Τελευταία ερώτηση. Τι κάνατε για τις εταιρικέ σχέσεις ασφαλείας και αυτή την περίπτωση την υπόθεση τρομοκρατίας σε συνεργασία με τους Γάλλους συναδέλφους για αυτή την υπόθεση τρομοκρατίας. Είναι μόνο μία υπόθεση που, είναι, που έχει ξεκινήσει για αυτά τα θέματα φέτος. Αλλά είναι ε, σημαντική γιατί αυτός ο ύποπτος τρομοκρατίας και που είχε τέτοιο πλωστάσιο και εκρηκτικά ξέρουμε ότι είχε διασυνδέσεις μεγάλους αστυνομικούς και με άλλα άτομα στη Γαλλία Ενημερώσαμε τους Γάλλους συναδέλφους για όλα τα στοιχεία που είχαμε και νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας. Βέβαια δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση, αυτό είναι σαφές. Όπως ξέρετε, σε τέτοιες υποθέσεις δεν είναι καλό να γράφουν πολλά εφημερίδες για να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η περίπτωση καθιστά σαφές σε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάνουμε προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και την τρομοκρατία που πολλές φορές ε, εκπορεύεται από το Κρεμλίνο. Τώρα αν μπορώ να πω δύο λόγια ως ε, πολίτης απλώς και όχι ως εισαγγελέας. Σας παρακαλώ να στηρίξετε τις προσπάθειές μας ε, για την απελευθέρωση της, ε, των θεωρήσεων. Όχι γιατί θα έρθουν τόσο πολλοί. Το 80% των πολιτών μας ε, ουδέποτε έχει επισκεφθεί την Ένωση. Και επειδή η οικονομική κατάσταση, η μισθή, η οικονομία μας έχουν πολλά προβλήματα, δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ένωση. Αλλά όλοι οι Ουκρανοί που ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα ανατολικά μας σύνορα είναι πολύ χρήσιμο να λάβουν αυτό το μήνυμα από τους ε, συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα να πάρουν ε, βίζα και διαβατήριο. Δεν είναι θέμα να επισκεφθούν ε, την Ένωση. Είναι θέμα να δουν την αλληλεγγύη σας και το γνωρίζω. Γιατί ξέρετε, ο γιος μου ήταν θελοντής στην πρώτη γραμμή των ε, μαχών κοντά στο αεροδρόμιο του Ντανιέτσκ. Ξέρω πολύ καλά πώς σκέφτονται οι στρατιώτες. Δεν θέλουν ε, βοήθεια σε τεχνικό επίπεδο. Θέλουν αλληλεγγύη. Γι' αυτό σας παρακαλώ δείξτε αυτήν την αλληλεγγύη της Ευρώπης στην κοινή μας προσπάθεια καταπολέμησης της βαρβαρότητας, της τρομοκρατίας αυτός είναι ο κοινό μας αντίπαλος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά τα πολύ συγκινητικά σας λόγια. Θα τα θυμόμαστε. Ε, ο κύριος Κένεθ Ντίν, αν θέλει να παρέμβει, έχετε το λόγο. Η κυρία Χάρμς επίσης ζήτησε το λόγο. Ε, ένα-δύο σχόλια για τα ερωτήματα που τέθηκαν. Όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτος. Και ένα από τα βασικά κριτήρια βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι Ουκρανικές αρχές είναι ε, ο σεβασμός ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως φίλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και επίσης άποψή μας είναι ότι η αστυνόμευση, η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης δεν αφορά μόνο την καταστολή, αλλά αντιθέτως τη χρήση των πιο ήπιων μέσων για τον έλεγχο και η χρήση βίας θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, μόνο με απολύτως νόμιμο τρόπο, όταν δεν υπάρχει καμία άλλη οδός για να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση. Η χρήση της βίας είναι τελευταίο καταφύγιο. Πάντοτε η συζήτηση είναι καλύτερη από τη βία. Και τέλος, ε, βοηθούμε στη διαφύλαξη των συνόρων και σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής μας είναι ακριβώς αυτό, να ενισχυθεί ε, η διασύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Άρα δεν ωφελείται μόνο η Ουκρανία από την αποστολή μας, αλλά και οι 28 χώρες της Ένωσης. Γιατί αποκτούμε διεθνείς δεσμούς και νομίζω ότι η όλη μας δραστηριότητα θα ενισχύσει και τις δικές μας ε, δυνατότητες, ικανότητες ε, καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ η κυρία Ρεμπέκα Χάιμς. Ναι, να πω κάτι προς υποστήριξη των όσων είπε ο κύριος Λουτσέγκο. Το Σαββατοκύριακο εγώ πραγματικά είδα πραγματική δυσαρέσκεια από ανθρώπους στο Κίεβο για τις νέες συζητήσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δεν το πιστεύουν. Πολλοί από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη συζήτηση που γίνεται εδώ δεν το πιστεύουν ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, διότι δεν πιστεύουν ότι ε, όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανακύψει σχετίζονται με τη δική τους πρόοδο, αλλά σχετίζονται με την Τουρκία. Τώρα ασκείται επιπλέον πίεση λόγω των εξελίξεων με τη Γεωργία. Δεύτερη δυσαρέσκεια σχετίζεται με, την, με τις κυρώσεις. Ξέρουν οι Ουκρανοί ότι δεν έχουν ληφθεί ε, στρατιωτικές κυρώσεις για την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι ενώ οι συγκρούσεις ε, αυξάνονται και τον τελευταίο μήνα σκοτώθηκαν 30 άνθρωποι στην Ανατολική Ουκρανία, από ευρωπαϊκής πλευράς αρχίζουν και εμφανίζονται φωνές ε, αμφισβήτησης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί ε, κατά της Ρωσίας. Και αυτό δεν βοηθάει το κλίμα υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Συμφωνώ. Φυσικά έχουμε αυτή τη συμμορία του Ιωαννούκοβιτς και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα δίκτυα, άλλες ομάδες μεγαλοκαρχαρίων και αυτοί βρίσκονται, έχουν διεισδύσει σε όλο το πολιτικό φάσμα. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαίοι θέλουμε κάποιος να τεθεί επικαφαλής του Γραφείου της Γενικής Εισαγγελίας που να είναι πολιτικά ανεξάρτητος. Και αυτό δεν αποτελεί μια αμφισβήτηση κατά ε, ημών με ύψιλον προσωπικά, αλλά αποτελεί ένα αίτημα για την απαραίτητη, την αναγκαία πολιτική ανεξαρτησία του Γενικού Εισαγγελία από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Διότι, όπως είπατε, τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει η αλλαγή αν για άλλη μια φορά ο Ουκρανικός λαός χάσει την εμπιστοσύνη του στο, στη διαδικασία εκδημοκρατισμού, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω να τονίσω για άλλη μια φορά την εξέχουσα σημασία που έχει η συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Ουκρανικής αστυνομίας γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους κοινού πολίτες να δουν οι άνθρωποι αυτοί ότι το κράτος τους προσφέρει ασφάλεια σε καθημερινό επίπεδο. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική και η εδαφική ακαιρεότητα και η διαφύλαξη των συνόρων και δεν θα το αμφισβητήσει κανένας Ουκρανός αυτό. Αλλά υπάρχει και αυτό, αυτή η κλίμακα η προσωπική της καθημερινής ζωής των ανθρώπων όπου και εκεί πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες προσπάθειες μεταρρύθμισης εξυγχρονισμού και νομίζω ότι το έργο σας και οι συνολικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα ίσως δεν έχουν αποφέρει ακόμα ε, ή μάλλον δεν αναδεικνύεται πολύ συχνά ως κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ όμως διαπίστωσα η μαλλον δεν αναδεικνυεται πολυ συχνα ως κατι πολυ σημαντικο εγω ομως διαπιστωσα η όμαση ε, για το σημαντικότατο έργο που έχετε κάνει και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Οι, οι, οι ιδιαίτερες μου, ε, τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου θα ήθελα να τις απευθύνω στον επικεφαλής της αποστολής. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καθόλου χρόνο. Ο Γενικός Εισαγγελέας ε, δυστυχώς πρέπει να φύγει ε, για το αεροδρόμιο. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά, κύριε Εισαγγελέα, κύριε Λατσίνσκας, κύριε Αντίν. Α, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω, λέει ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, για την ευχαριστή για την δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω εδώ να κάνουμε αυτή την εξαιρετικά ποιοτική συζήτηση. Να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή Ντίν και τον κύριο Λαντσίνσκας για την αποστολή. Ελπίζουμε η αποστολή αυτή να συνεχίσει να μας παρέχει την βοήθειά της, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο επιθεμείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much indeed.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 επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο αλλά ελπίζω το επόμενο θέμα να είναι εξίσου ενδιαφέρον. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω την δραστηριότητα της EU Pol στο Αφγανιστάν. Επιτεύγματα προκλήσεις και προοπτικές πέραν του 2016. Καλωσορίζω λοιπόν τους προσκεκλημένους μας σήμερα, την κυρία Πία Χέρνβαλ ελπίζω να είπα το όνομα σας σωστά λέει πρόεδρος, Σκολούτσι Κολυγάκη, που συνοδεύεται από το γνωστό μας και ενευθύν το διευθυντή στο CPCC στην ΕΕΔ. τέλος του τρέχοντος έτους θα λήξει και η εντολή της EUPOL της αποστολής δηλαδή που βρίσκεται στο, στο Αφγανιστάν από το 2007 και θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρη απολογισμό των επιτευμάτων αυτής της αποστολής. Γι' αυτό ακριβώ θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή μα για αυτό το σκοπό. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Τιν, στον διευθυντή, και μετά στην κυρία Πία Βαλ, που είναι επικεφαλής αποστολής, αν θυμάμαι καλά. Θα δώσω το λόγο πρώτα λοιπόν στον κύριο Κενευτίν. Παρακαλώ. Κύριε Ντίν. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την κυρία Στένβαλ που ηγήθηκε αυτής της αποστολής με πολύ επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Όπως ξέρετε θα εκπνεύσει η εντολή στο τέλος του έτους. Ήταν περιβάλλον που αποτελούσε πρόκληση η δράση αυτή στο Αφγανιστάν. Εκτιμώ λοιπόν την δράση τη και την συγχαίρω όπω και τα υπόλοιπα μέλη τη Αποστολή, για αυτά που πέτυχαν υπό συνθήκες αντίξωε. Θα συνεχίσει λοιπόν να κάνει ό,τι μπορεί η αποστολή μέχρι το τέλο τη εντολή τη, για να βοηθήσει το λαό και τις αρχές του Αφγανιστάν να είναι πιο αξιόπιστες πιο αμερόληπτες επίσης όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου στην Καμπούλ και στις υπόλοιπες επαρχίες της χώρας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πια. Συγχαρητήρια σας και στους συναδέλφους σου. Παρακολουθώ την πορεία της αποστολής τα τελευταία 9 χρόνια και πρέπει να πω ότι θα μπορούσε κανεί να ασκήσει ενδεχομένω σωστά κριτική για κάποια πράγματα που μπορούσε να έχει κάνει η αποστολή. Έχουμε όμως μια θετική στάση ω απολογισμό για το τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι έγινε, τι δεν έγινε και υπενθυμίζω ότι ήταν αρκετά περίπλοκη και ασταθής η κατάσταση. Κατά διάρκεια της μεγαλύτερης περίοδου της Πάντως να σας πω ότι η αποστολή είχε σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά την ε, βοήθεια στην αστυνομία, στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βέβαια ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει την σύστασή τους, αλλά βοήθησε πάρα πολύ η αποστολή στην παροχή αστυνομικών υπηρεσιών όπου δεν υπήρχαν. Και αυτό βοήθησε βεβαίως την κυβέρνηση στην καταπολέμηση των Ταλιμπάν και των εξτρεμιστών. Αλλά από τη στιγμή που η κατάσταση ήταν αυτή που ήταν στο Αφγανιστάν όσον αφορά την αστυνόμευση, νομίζω ότι οι επιτυχίες μας ήταν σημαντικές και τουλάχιστον τώρα η κυβέρνηση κατανοεί την σημασία ύπαρξης μιας αστυνομικής δύναμης. Πολιτοφυλακής ενδεχομένω, που δεν σημαίνει βέβαια μια υποδέστερη αστυνόμευση, αλλά σημαίνει βέβαια αστυνόμευση μέσω της ε, πυθού και μια μορφή αστυνόμευσης που μπορεί ο κόσμος να εμπιστεύεται και να λύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αυτή λοιπόν η αστυνομική, αστική μάλλον αστυνομία, η πολιτική αστυνομία, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να υπάρχει και να έδωσε βέβαια επιτήρησης από την κυβέρνηση για αυτή τη μορφή αστυνόμευσης Αν δούμε σε άλλες χώρες, έχουμε μια τέτοια μορφή αστυνόμευση, η οποία υποστηρίζεται από πιο στρατιωτικές μορφές αστυνόμευσης. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να αποδεχτεί το γεγονός ότι αυτή η αστική αστυνομία έχει σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει βέβαια τα θέματα που είναι φλέγοντα, αλλά βεβαίως για το κράτος δικαίου έχουν τεράστια σημασία οι μα. Είχαμε συνεργασία των διαφόρων Υπουργείων και Αρχών, Υπουργείο Δικαιοσύνη, ώστε να υπάρξει τελικά μια κατάλληλη νομοθεσία, χωρίς την οποία βέβαια δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για την αστυνόμευση. Οπότε νομίζω ότι η αποστολή ήταν αρκετά επιτυχή από αυτή τη σκοπιά και μπόρεσε να κάνει ένα capacity building στα πλαίσια των Υπουργείων, σε συνεργασία με υπουργού, υφυπουργού και τον ίδιο τον πρόεδρο, ώστε να περάσει αυτή η νοοτροπία που ανέφερα προηγουμένω. Πάντω, Πρόεδρε, μετά το 2016 θα πρέπει οι χώρες μίλη να εξετάσουν τη μορφή παρουσίας της αποστολής αλλά θα πρέπει να δούμε λοιπόν το Γενάρη ακριβώς ποια θα είναι ακριβή μορφή της παρουσίας σε τι θα εστιάσει η αποστολή Αυτά. Θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πία Στιένβαλ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για την αποστολή μας στην Καμπούλ, στο Αφγανιστάν. Θα επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα, σύντομα. Καταρχάς το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε η οικονομική, η πολιτική και η κατάσταση ασφαλεία στη χώρα. Θα μιλήσω για τα επιτεύγματα κατά δεύτερο λόγο των δύο τελευταίων ετών και που βρισκόμαστε τώρα. Και τρίτον, κάποια συμπεράσματα και διδάγματα. Η πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι πολύ ασταθής. Όπως ξέρετε έχουμε μια κυβέρνηση εθνική ενότητας που αποτελείται από τον Προδεκάνη και τον κύριο Απτούλα. Ήταν δύσκολο για αυτούς λοιπόν να λάβουν αποφάσεις και να πετύχουν ακόμα και τους διορισμούς των Υπουργών. Κατά διάρκεια παρουσία μα είδαμε 8 υπουργού και ο νέος υπουργό είναι στρατιωτικός. Αλλά φαίνεται να είναι καλό. ή τουλάχιστον λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά και γρήγορα, οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτόν. Στο Αφγανιστάν επίση υπάρχει σημαντική αμερικανική επιρροή η οποία επηρεάζει και τη δική μας τη δουλειά επειδή οι Αμερικανοί είναι υπέρ της αστυνόμευσης όταν υπάρχουν μόνο εξεργέσεις ή κατά των ναρκωτικών για τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει η στρατιωτική αστυνόμευση και ο πρόεδρος κάνει παίρνει πολλές αποφάσεις μετά από Συμβουλέ ε, των Αμερικανών για τα στρατιωτικά και όχι για τα αστυνομικά θέματα. Η φτώχεια έχει αυξηθεί από πέρσι. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν θέσει εργασία, δεν υπάρχουν επενδύσει. Ο κόσμο έχει απελπιστεί. Και είναι κύριο λόγο αυτό για τη μετανάστευση. Γι' αυτό ακριβώ οι γενιέ που σπούδαζαν και είναι πτυχιούχοι αποφάσισαν να φύγουν, να πάνε στην Ευρώπη και πολλοί από αυτούς τους νέους που έρχονται εδώ, δηλαδή στην Υπηρώ μας. Είχαμε και αυτό το μεταβατικό σχέδιο για την οικονομική αλλαγή και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί και ακόμα δεν έχουμε πετύχει την ανάκαμψη της οικονομίας. Η οικονομική λοιπόν κατάσταση δεν είναι και αυτή καλή. Για την ασφάλεια τώρα, η κατάσταση είναι ενδιαφέρουσα. Στην Καμπούλ η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί σχέση με πέρσι. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε επαρχία υπάρχουν μάχες. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακριβώ ποια είναι η πραγματική κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα. Έχουμε πολλούς Ταλιμπάν και κάποιους μαχητές του ISIS. Και υπάρχει απόκληση απόψεων κατά πόσο είναι παρόν το ISIS, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η κατάσταση για την ασφάλεια, η οποία θα λέω το λιγότερο δεν είναι καλή. Μια και έχουμε και νέο ηγέτη για του Ταλιμπάν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο μέλλον. Αυτή είναι λοιπόν κυρίως η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Να σας πω και δύο λόγια για την αποστολή. Έχουμε 130 άτομα διεθνέ προσωπικό και άλλα τόσα Αφγανούς. Πάντοτε ταξιδεύουμε με θωρακισμένα αρχήματα b B6 με συνοδεία ασφαλείας στις μετακινήσεις μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Να περάσω τώρα στα δύο τελευταία χρόνια. Τι έχει γίνει. Επικεντρωθήκαμε όχι μόνο στη βασική μας εντολή, αλλά και στις δράσεις μας που βασίζονται στο γεγονό ότι αν διαφωνούν οι θύνοντες, τότε θα πρέπει να κάνουν δουλειά με τους πολίτες. Πριν δύο εβδομάδες δώσαμε στον κύριο Απτουλά 11 συστάσεις για αλλαγές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτός υποσχέθηκε να κάνει μια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για να, δούμε, για να δούνε πώς μπορούν να προωθήσουν αυτές τις συστάσεις. Αυτό πριν δύο χρόνια δεν θα μπορούσε να συμβεί. Οπότε είναι καλό τώρα που δείχνουν κάποιο έτσι ενδιαφέρον για την ύπαρξη έτσι αστυνομίας πολιτών πέραν των αστυνομικών δηλαδή των συγγνώμη των στρατιωτικών υπάρχει λοιπόν μια αποδοχή μια θετική κατανόηση των θέσεών μας είχαμε επίση μια συνάντηση με την Ουλακάν με την σύζυγο του Πρόεδρου που ενδιαφέρεται για το θέμα της αστυνομίας, της πολιτικής αστυνομίας Είπαμε να κάνουμε δύο σεμινάρια στην Καμπούλη για αυτό το θέμα και το θέμα της εθνικής αστυνομίας στο Αφγανιστάν ήταν προβληματικό γιατί όλοι έχουν διαφορετική αντίληψη για το τι θα πρέπει να είναι η αστυνόμεση στο Αφγανιστάν. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσω των δρασεών μας να προωθήσουμε ακριβώς τη σύσταση αστυνομία με πολίτε, το τι θα πρέπει να κάνει, τι αρμοδιότητε θα έχει κτλ. Μιλήσαμε επίση και με τον κύριο Απτουλά και με τον πρόεδρο για τα θέματα ασφαλεία. Αν δούμε, α πούμε, το θέμα τη νομοθεσία για την αστυνομία και το στρατό και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλεία δεν έχουν διαχωρισμό αρμοδιοτήτων. Οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να συνεργαστούν. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Επίσης, να σας πω δύο λόγια για τα επιτεύγματά μας. Αυτά που είπε και ο Κέν προηγουμένως για την συγκρότηση αστυνομίας πολιτικής. Όταν ήρθα το 2010 σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι βέβαια πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά δυστυχώ η κατάσταση, ιδιαίτερα σαν αφορά την ασφάλεια, έχει επιδεινωθεί. Το 7, όταν ξεκίνησε η αποστολή, υπήρχαν προσδοκίε ότι εντωμεταξύ η πολιτική αστυνομία θα ήταν η κύρια μορφή αστυνομεύση στο Αφγανιστάν. Αυτό δεν έχει γίνει, αλλά τώρα έχουν τη γνώση, φαίνεται να έχουν και την βούληση, οπότε αυτό είναι επίτευγμα. Επίσης να σας πω ότι έχουν και ένα σχέδιο για τις γυναίκες στο Υπουργείο όσον αφορά την αστυνομία, ώστε το περιβάλλον για τις γυναίκες αστυνομικούς να είναι καλύτερο και να υπάρχουν ψηλότεροι αριθμοί τους. Ε, έχουμε 5.000 γυναίκες και ε, θα, ε, ως το έχουμε 5.000 και αν μένουμε 10. Προς το παρόν έχουμε 3.000. Αν όμως δεν υπάρχει και το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τις γυναίκες δεν θα έχουμε επαρκέ αριθμούς. Επικεντρώμαστε λοιπόν στις γυναίκες ώστε να υπάρχουν κατάλληλες δυνατότητε για αυτές να δουλέψουν. Η Αστυνομική Ακαδημία επίσης. Άλλο ένα θέμα που συζητάμε με το Υπουργείο Εσωτερικών Επίσης οι εκπαιδευτές των Ακαδημιών. Το 14, ήδη από το 14, δημιουργήσαμε μια Ακαδημία μόνο για Αυγανούς και συμβουλέψαμε τους επικεφαλείς και νομίζω ότι τα κάνουν πια μόνοι τους, τα καταφέρνουν μόνοι τους και πάει καλά. Ο Υπουργός θέλει τώρα να έχουμε και μεταπτυχιακά, μάστερ, για αυτές τις σχολές και νομίζω τα πράγματα πάνε καλά. Επίσης πριν δύο εβδομάδες έχουμε και το δημοσιολαβητή, τον αστυνομικό. Θα υπάρχει λοιπόν ένας δημοσιολαβητής για την αστυνομία. Και θα έχουμε διαδικασίες που θα αφορούν και τους και τις αστυνομικές δράσεις αλλά ο αστυνομικός εισαγγελέας βέβαια θα πρέπει να συνεργάζεται ώστε να έχουμε καλύτερη διεκπαιρέωση των διαφορών υποθέσεων. Επίσης, πρέπει να δούμε και τα θέματα διαφθοράς. Και να σας πω τέλος ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαφθοράς, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια της αποστολής. Αλλά δεν αφορά μόνο τη δικιά μας αποστολή ή την αστυνομία. Αν δεν αντιμετωπίσουμε σφαιρικά την διαφθορά στο Αφγανιστάν, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και βιώσιμη ειρήνη στο Αφγανιστάν δεν θα υπάρξει αν δεν συγκροτηθεί πολιτική αστυνομία. Αυτά είχα να σας πω Ευχαριστώ να απαντήσω βέβαια και σε ερωτήσει σα για να καταλάβετε καλύτερα το τι κάνουμε εκεί. Ευχαριστώ. Βεβαίω και θα σα κάνουμε πολλέ ερωτήσει, λέει ο Πρόεδρο. Είναι ο παρόν ο κύριο Πέτρα Οστεβίτσο που είναι ο επικεφαλή τη αντιπροσωπή για σχέση με το Αφγανιστάν. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Να εκφράσω την εκτίμησή μου για τι προσπάθειέ μα τη επικεφαλή τη Ιού Πόλη του Αφγανιστάν. Είναι πολύ απαιτητικά τα καθήκοντα χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια για να μπορέσετε να εκτελέσετε τα καθήκοντά σας παντού στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αφοσίωσή σας. Πρώτον, να ασχοληθώ με την εντολή σας, τα καθήκοντά σας. Να γίνει υψηλότερος ο βαθμός του επαγγελματισμού της αστυνομίας του Αφγανιστάν, να υπάρξει κατάρτιση και να βελτιωθούν και οι διοικητικές δυνατότητες. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε για να βοηθήσετε την αστυνομία του Αφγανιστάν να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις. Χρηματοδότηση. Προσλήψεις των καταλήλων ε, αστυνομικών. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ λίγο περισσότερα για το πώς λειτουργεί η αστυνομία και άλλοι θεσμοί στις διάφορες περιοχές της χώρας γιατί βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή αστυνομία στην Καμπούλ και τα περίχωρα αλλά ξέρουμε ότι το Αφγανιστάν είναι τόσο μεγάλη χώρα με τόσο μεγάλες ε, ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή. Από περιοχή σε περιοχή είναι εντελώ διαφορετική κατάσταση. Και τέλος, ε, έχω εκτίμηση μεγάλη για τις προσπάθειές σας ε, στο παρελθόν και το παρόν, αλλά τι θα γίνει μετά το 2016. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα μαζέψουμε το Δεκέμβρη. Με βάση την πείρα σας, πόσο καιρό ακόμη και τι προσπάθειες πρέπει να κάνουμε τα επόμενα έτη. Βεβαίω θέλουμε συνεργασία και έχετε την πλήρη στήριξη τη αντιπροσωπεία μα. Κατανοώ την σημασία τη αποστολή σα και ε, με, είμαι πολύ ικανοποιημένο από αυτή τη δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ανούντα Οζόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σα. Σα συγχαίρω για την εργασία σας. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η αποστολή σας. Ε, μας το επενθυμίσατε. Σας επισκέφθηκα δύο φορές υπό διαφορετικές ιδιότητες και σας ομολογώ ότι έχω ακόμη πολλά ερωτήματα για το τι πάμε να κάνουμε εκεί πέρα. Ε, βεβαίως ε, να μην υπάρχει παρανόηση, δεν θέτω ένα αμφιβόλο το υψηλό επίπεδο και την ε, ευσυνειδησία των παρόντων εκεί. Ξέρω πόσο δύσκολες οι συνθήκες εργασίας και επιτελούν τα καθήκοντά τους με πολλή ευσυνειδησία. Αλλά ποιος είναι ο στόχος μας δεν είναι πολύ σαφής ε, σε μένα τουλάχιστον. Είπατε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον ασφαλείας ιδιαίτερα κακό όπου το θέμα δεν είναι να καταρτήσουμε γυναίκες αστυνομικούς αλλά να αντιμετωπίσουμε μία ένοπλη εξέγερση και τρομοκρατία. Οπότε οι προτεραιότητες οι δικές μας με βάση την αρχική εντολή δεν είναι οι προτεραιότητες των ίδιων των Αφγανών. Θυμάμαι πολύ καλά τις συζητήσεις που είχαμε στην προηγούμενη επίσκεψή μας στην Καμπούλ όπου ο επικεφαλής της αστυνομίας της Καμπούλ ε, χαιρόταν ιδιαίτερα που είχε Ευρωπαίους αστυνομικούς παρόντες και μας είπε όμως, ξέρετε τώρα, εμάς αυτό μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πόσους Ταλιμπάν έχουμε μεταξύ των αστυνομικών στα αστυνομικά μας τμήματα και πότε θα αρχίσουν να μας σκοτώνουν. Τώρα αυτά τα θέματα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας λέτε τι κάνετε στη Δύση, αλλά άλλα προβλήματα έχουμε. Δηλαδή, τον τρόπο εργασία μας, τις προδιαγραφές μας, τα πρότυπά μα δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Άρα είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Εννιά χρόνια έχουμε αυτή την αποστολή στο Αφγανιστάν και κάνουμε ακόμη συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τον τρόπο λειτουργίας του. Μα, καλό αυτό, αλλά παίζουμε κανένα ουσιώδη ρόλο σε σχέση και με το προσωπικό που χρησιμοποιούμε, με τους στόχους που έχουμε, η ΕΠΟΛ μπορεί να παίξει ουσιώδη ρόλο, να έχει ουσιαστική και μακροπρόθεσμη επίπτωση. Είναι μια ερώτηση. Εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες, αλλά παρόλα αυτά είναι ερώτηση. Δεύτερον, όπως είπατε, τι σημαίνει αστυνόμευση στο Αφγανιστάν με βάση την κατάσταση, το παρελθόν. Ε, πολύ περισσότερο είναι στρατιωτικός ο ρόλος της αστυνομίας. Δηλαδή πρέπει να ασχολείται και αυτή με την καταπολέμηση της εξέγερσης. Δεν είναι αυτός ο κλασικός ρόλος μιας αστυνομίας. Οπότε πρώτο ρόλο παίζουν άλλοι εταίροι. Πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι περιφερειακοί, παγκόσμιοι, πολυμερείς, που επίσης παρεμβαίνουν. Θεωρείται λοιπόν ότι ο τρόπος παρουσίας μας και η θέση που κατέχουμε σε σχέση με αυτούς τους άλλους εταίρους μας επιτρέπει να παίξουμε ουσιώδη ρόλο που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Αφγανών. Αυτά. Αλλά και κάτι άλλο, κάπως δευτερεύον μία ερώτηση που θέτω σε όλους τους επικεφαλείς ε, των αποστολών μας, των αντιπροσωπιών μας, όπου έχουμε αποστολές ε, συμβουλών και κατάρτισης, οι επιτόπου, εκεί οι χώρες που λαμβάνουν και οι αρμόδιοι τους μας λένε όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, σας ευχαριστούμε. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να μας δίνετε συμβουλές, αλλά και εξοπλισμό. Ξέρω τώρα τους περιορισμούς ε, που έχει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και οι επικεφαλής των αποστολών έχουν ακόμη λιγότερη αυτονομία. Λαμβάνετε τέτοια αιτήματα από τους Αφγανούς και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Αναγκόμες. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι εδώ νωρίτερα και να ακούσω την παρουσίασή σας. Πήγα στο Αφγανιστάν το 2008, μόλις είχε δημιουργηθεί δηλαδή η αποστολή μας, η UPOL, και τότε ε, πράγματι είχε αποτελέσει μεγάλη πρόοδο το γεγονός αυτό. Με είχε εντυπωσιάσει τότε το γεγονός ότι είχαμε μάθει ότι Περισσότερες, περισσότεροι από τους μισούς κρατούμενους στο Αφγανιστάν τότε ήταν γυναίκες, οι δεν είχαν κάνει τίποτα, δεν είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα, αλλά το μόνο που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να ξεφύγουν από οικογένειες και συζύγους που τις κακοποιούσαν. Αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση, σε ποιο βαθμό έχετε καταφέρει να συμβάλλετε στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι γυναίκες έχουν πάψει να αποτελούν την πλειονότητα των κρατωμένων. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε πλέον γυναίκες αστυνομικούς έχει συμβάλει στο να αλλάξει η κατάσταση. Και φυσικά το θέμα αυτό δεν συνδέεται μόνο με την αστυνομία αλλά και με τη δικαστική εξουσία η οποία δεν ήταν ανεξάρτητη, ήταν ε, πλήρως διεφθαρμένη, δεν παρουσίαζε καμία ηθική ακαιρεότητα και καθοδηγούνταν από εντελώς εσφαλμένα κίνητρα. Έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση. Όταν ε, ε, επισκέφτηκα πρόσφατα την Ελλάδα, είδα σε καταβλητισμούς προσφύγων πάρα πολλές γυναίκες. Κάποιες με τα παιδιά τους, άλλες ήταν μόνες τους. Δεν συνδέεται και αυτό με την κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες στο Αφγανιστάν, στο για πολιτιστικούς αλλά και για άλλους λόγους. Η κυρία Λόζιν, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ε, στα όσα είπε και η κυρία Γκόμες. Γνωρίζω και εγώ αυτήν την έκθεση. Άκουσα όμως ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στη φυλακή παρά εκτός φυλακής. Αυτό βέβαια δεν κάνει την κατάσταση καλύτερη. Το αντίθετο, χειρότερη την κάνει. Απλά ήθελα να συμπληρώσω και αυτό το στοιχείο. Μετά, έχω ερωτήματα για, το κόστος. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος των ε, ενόπλων δυνάμεων του ε, Αφγανιστάν. Άλλοι μιλούν για 4 δισεκατομμύρια ε, δολάρια, άλλοι για 6 δισεκατομμύρια κατέτος. Αυτή, η εκτίμηση αφορά την, ε, την μείωση κατά 230.000 του προσωπικού των ε, ενόπλων δυνάμεων που είχε αποφασιστεί το 2016 αλλά που τελικά ανεκλήθη. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του, του Broking Institute, το 2015 σκοτώθηκαν 7.000 ε, άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας σε συγκρούσεις ε, είναι υπερβολικά, υψηλά, ε, υπερβολικά υψηλή αυτή η αριθμή. Επίσης, οι ΙΠΑ δίνουν 60% της ανθρωπιστικής τους βοήθειας για την ανάπτυξη του τομέα ασφαλείας ε, στο Αφγανιστάν. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο είναι. Επίσης, η αποστολή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί μη στρατιωτική πολιτική ή μήπω είναι στρατιωτική ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αλληλοδιαπλοκή μεταξύ αστυνομία και στρατού. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Στετίνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ για τα στοιχεία που μας δώσατε για τις αστυνομικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί ε, εγώ έζησα δυόμιση χρόνια στο Αφγανιστάν και ασχολήθηκα με την εκπαίδευση των αστυνομικών ε, δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό και το ερώτημά μου το ISAF αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί πολλοί από τους αστυνομικούς που είχαν εκπαιδευτεί έφυγαν, ε, λιποτάκτησαν γιατί πολλοί φύλαρχοι ε, και τοπικοί ηγέτες τους ε, πρόσφεραν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι, έχετε συνεργασία με μονάδες της ISAF και του ΝΑΤΟ και αν ναι, ποια μορφή ε, είχε αυτή η συνεργασία. Ωραία. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την συμμετοχή της ΙΟΥΠΟ όσον αφορά τη συμβολή της όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών και ποια είναι η εμπειρία σας ε, μέσω της συνεργασίας σας με τη Europol. Δεύτερον, από τις συζητήσεις που έχω κάνει με μέλη των αστυνομικών δυνάμεων από διάφορες χώρες ε, και από την Πολωνία και από την ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία οι οποίοι είχαν βρεθεί στο Αφγανιστάν μπορώ να σας πω ότι Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που ε, ε, απέφερε στην κεντροαφρικανική δημοκρατία ε, η εκεί αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η δυνατότητα που είχαν οι αστυνομικοί που έκαναν τις περιπολίες να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Ήταν η, η εμπειρία που είχαν αποκομίσει από το Αφγανιστάν. Το, το ερώτημά μου συνδέεται με την παρέμβαση του κ. Νταζάντ. Ότι πιθανότατα και κάπως το επενηθήκατε κι εσείς ότι ότι η στρατιωτική αστυνομία, οι στρατιωτικές περιπολίες είναι απαραίτητε λόγω της πολύ τεταμένη κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα και τι διαδικασίες έχετε εφαρμόσει για να ενισχύσετε τη δική σας θέση και την δική σας συμβολή και το προφίλ πολιτικής αστυνομίας που εσείς θέλετε να στηρίξετε. Και τέλος, για τη μετανάστευση ένα ερώτημα. Έχετε στοιχεία να μας δώσετε. Ποια είναι η έκταση της μετανάστευσης ανθρώπων προς την Ευρώπη. Αναφέρθηκε ένας αριθμός γυναικών, αλλά είναι βέβαιο ότι το τωρινό κύμα προσφύγων που δέχεται η Ευρώπη δεν αποτελείται αποκλειστικά από ανθρώπους που προέρχονται από τη Συρία αλλά και από ανθρώπους που προέρχονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με αυτές τις προσφυγικές ροές Κύριε Ντίν και κυρία Στενουάλ. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να τις σημείωσα όλες. Αν δεν τα καταφέρω να απαντήσω σε όλες, είμαι στην διάθεσή σας. Για την, ε, για, τις, την κατάρτιση και την επαγγελματικοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Ε, ρωτήσατε ποιος Ποιε είναι οι προκλήσει. Μισθός του αστυνομικού στην Καμπούλ είναι 150 δολάρια. Το ενίκιο όμως για ένα διαμέρισμα είναι 300 δολάρια. Άρα οι άνθρωποι αυτοί εξαναγκάζονται να διαφθαρούν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Η διαφθορά λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεύτερο θέμα είναι ε, οι προσλήψεις και η στρατολόγηση με βάση τις ικανότητες. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Στο Αφγανιστάν οι περισσότερες οικογένειες ε, έχουν σχέσεις μεταξύ τους και αν δεν έχεις συγγενή ε, δεν μπορείς να βρεις λύση στο πρόβλημά σου ή να βρεις κάποια θέση. Προσπαθούμε να να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και όσον αφορά την πρόσληψη ανθρώπων για την ΆΜΠΑ, την, την Αστυνομική ε, Ακαδημία, αλλά και για την ίδια την αστυνομία, τις αστυνομικές δυνάμεις και τη στελέχωσή τους. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να παρέχουμε στρατηγικού χαρακτήρα σύμβουλε. Δεν κάνουμε κατάρτιση, αλλά προσπαθούμε να αλλάξουμε την οτροπία αυτών των ανθρώπων. Προσπαθούμε να του κάνουμε να καταλάβουν γιατί θα του ωφελήσει του ίδιου να κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Γιατί θα του βοηθήσει και του ίδιου και θα του ωφελήσει και του ίδιου να γίνονται προσλήψει με βάση τι ε, ικανότητε των ανθρώπων, των υποψηφίων. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν και γυναίκε μέσα στην αστυνομία και ε, νομίζω ότι αν αλλάξουμε ακόμα και την νοοτροπία ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε υψηλή θέση θα έχουμε κάνει κάτι. Φυσικά οι στόχοι μας είναι μεγαλύτεροι, αλλά και αυτό κάτι θα είναι. Δεύτερο ερώτημα για την αποστολή μας. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει ε, πολιτική αστυνομία στο Αφγανιστάν θα υπάρξει και ειρήνη. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ ανησυχώ για αυτό το ζήτημα. Ε, ε, γιατί σκοτώνουμε πάντοτε τους τροποκράτες. Γιατί δεν τους συλλαμβάνουμε, γιατί δεν τους βάζουμε στη φυλακή, γιατί δεν τους δικάζουμε. Γιατί γίνεται αποδεκτή αυτή η στάση απέναντι στους τρομοκράτες. Αν έχεις αστυνομικό, αστυνομική δύναμη η οποία ε, ε, αστυνομικό ο οποίος έχει καταλάβει, έχει πάει στην ακαδημία του, γνωρίζει τις αρχές του κράτους δικαίου, θα γνωρίζει πολύ καλά πώς να προστατευτεί, πώς να προστατεύσει και τον συλλαμβανόμενο και θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσει την ε, κοινωνία του και να εξασφαλίσει την ειρήνη στο, στη χώρα, στο Αφγανιστάν. Και όταν μιλάμε για στρατιωτική ε, αστυνόμευση, δεν μιλάμε ακριβώς για αυτό που ενδεχομένως φαντάζεται κανείς. Μιλάμε ε, για, για αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες πραγματικά ε, εισέρχονται στη μάχη. Και στις ε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κυκλοφορούν αστυνομικοί. Γιατί οι αστυνομικοί τελικά έχουν να υπομιστούν πολύ σοβαρότερες καταστάσεις και αντιμετωπίζουν πολύ δυσκολότερα, δυσκολότερες καταστάσεις από ό,τι πολλές φορές ο στρατός. Αν δείτε όμως την κατάσταση ε, σε σχέση με το 2001 ε, ίσως ε, δεν, ε, δεν, δεν υπάρχει βελτίωση που θα περίμενε κανείς. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Δεν είναι δυνατόν να εκπαιδεύουμε ανθρώπους και να σκοτώνουμε τους τρομοκράτες μόνο. About all of, about that. Um... Uh, λοιπόν, τα θέματα πώς θα πάει η αστυνομία στις διάφορες επαρχίες. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους Αφγανούς, ούτως ώστε τουλάχιστον οι επικεφαλείς των αστυνομιών στις διάφορες επαρχίες να έρχονται στην Καμπούλ για να ανταλλάσσουν ιδέες με το Υπουργείο και επίσης παρακολουθούμε πώς εφαρμόζονται οι κατευθυντήρες γραμμές του Υπουργείου Εσωτερικών στις επαρχίες. Γιατί δεν εφαρμόζονται πάντα και πρέπει να πω ότι οι εταίροι μας, GPPT που είναι Γερμανία αστυνομική, έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να παρακολουθήσουν αυτήν την ε, συμμόρφωση προς τις οδηγίες. Οι τοπικές αστυνομίες ε, μειώθηκαν από τις 130 στις 30, άρα αυτό ήταν θετικό γιατί χρειάζεται να παρακολουθήσουμε λιγότερες ε, αστυνομικές δυνάμεις. Ορισμένες φορές ε, δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι χαόδης η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Αλλά άμα έχει σωστό σχέδιο και αρχίζει σιγά σιγά να το εφαρμόζει με μικρά βήματα, μπορεί να επιτύχει ε, ουσιώδη αποτελέσματα. Σιγά σιγά. Και διάφορα άτομα που έχουν θετικές ιδέες, διάφοροι διοικητές, διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες, ε, επιτυχάνουν αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στο παρελθόν ήταν αδύνατο να μιλήσουμε με την αστυνομία για θέματα των καταναγκαστικών γάμων ανηλίκων, των παιδικών γάμων. Και φέτος το συζητήσαμε και φτιάξαμε κάποια βίντεο για την αστυνομία και φέτος μας υποσχέθηκαν ότι θα τα παίξουν στην εθνική τηλεόραση. Σε τηλεόραση που έχει εμβέλεια σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που μπορείς να επιτύχεις εάν έχεις μετροπαθεί ε, στόχους, μικρούς στόχους και τους εφαρμόζεις σταδιακά. Ε, λέτε ότι μπορεί να θέλουν και εξοπλισμό. Φυσικά μας ζητάνε συχνά εξοπλισμό γιατί τους αρέσει ο εξοπλισμός. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο λαό. Όμως η υπηρεσία μας ε, έχει προϋπολογισμό προγραμμάτων μόνο 400.000 ευρώ. Άρα δεν τους δίνουμε εξοπλισμό. Για τέτοια ζητήματα είναι το ΝΑΤΟ επιτόπου. Συνεργαζόμεθα με το ΝΑΤΟ. Αυτοί τους δίνουν ε, πολύ υλικό, αλλά εμείς όχι. Για ορισμένα προγράμματα που εφαρμόσαμε μπορεί να περιέχουν και κάποια μικρά στοιχεία υλικού, δηλαδή κάμερες για επίβλεψη μερικά τέτοια στοιχεία υλικού, αλλά σε μικρή κλίμακα. Κάτι που έχει αλλάξει από το 2010 όταν εργαζόμουν στην ε, Φινλανδέζικη Πρεσβεία. Τώρα συνεργαζόμαστε με όλους τους άλλους, με, δι... με διάφορες άλλες υπηρεσίες, το... την υπηρεσία Resolute Support, το SSMI που στηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, το GPPT, το UNAMA, το BNUNDP, το 2010 δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε τη στήριξη που δίνουμε στην αστυνομία, αλλά τώρα τη διαπιστώνω. Και είναι καλό που έχουν αυτή τη στήριξη. Και καλό είναι να υπάρξει και αυτή η χωροφυλακή, η gendarmerie, γιατί έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Και είναι χρήσιμο να ακούμε και διαφορετικές απόψεις και εμείς. Ίσως από αυτή τη διάσκεψη που θα κάνουμε τον Αύγουστο θα δούμε τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε στο μέλλον για να βοηθήσουμε την αστυνομία. Αυτοί δεν έχουν την ίδια δομή με την αφγανική αστυνομία. Και επίσης η συνεργασία μας με αυτή την υπηρεσία Resolute Support, αποφασιστική στήριξη, επίσης μας έχει βοηθήσει γιατί έχουν μια πιο στρατιωτική προσέγγιση για τις γυναίκες στις φυλακές. Ναι, υπάρχουν πολλές γυναίκες στις φυλακές. Που δεν έχουν καταδικαστεί. Τώρα όμως η Ρούλα κάνει, η γυναίκα του Πρόεδρου, γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις γυναικών στις αφγανικές φυλακές για να δούνε για ποιο λόγο κρατούνται. Χρειάζεται να παραμείνουν εκεί έχουν καταδικαστεί για κάτι ή απλώς κρατούνται χωρίς λόγο. Ορισμένες φορές καταλαβαίνω ότι είναι καλύτερα να είσαι μέσα παρά έξω από τη φυλακή γιατί μπορεί να έρθουν οι συγγενείς σου να σε δολοφονήσουν. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι χώροι όπου μπορούν, κάποιοι ασφαλείς χώροι όπου μπορούν να πάνε οι γυναίκες κάποια καταφύγια, αλλά δεν είναι και τόσο ασφαλή, ιδίω ε, αν έχει και παιδιά. Αν είσαι μια γυναίκα μόνη με παιδιά, είναι πολύ δύσκολο να βρει τα 5.000 δολάρια που χρειάζονται για να καταλήψεις τη χώρα. Πρέπει κάποιος να τους ε, στηρίξει άμα είναι να έρθουν εδώ. Τώρα για το κόστος, τα στοιχεία κόστους, δεν έχω ασφαλή στοιχεία. Ίσως δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις άμα σας δώσω στοιχεία. το οργανόγραμμα της Αφγανικής Αστυνομίας είναι 157.000, αλλά δεν νομίζω ότι όλες οι θέσεις έχουν καλυφθεί. Α, πόσο προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του, της διακίνησης ναρκωτικών. Δεν είναι στα πλαίσια της εντολής μας κάτι τέτοιο. Το μόνο που κάνουμε είναι, είναι ότι συμμετέχουμε σε διάφορες συναντήσεις για να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει και στηρίζουμε την Ίντερπολ σε μεγάλο βαθμό στο Αφγανιστάν. προσπαθούμε να λειτουργεί με πιο επαγγελματικό τρόπο το τμήμα της αστυνομίας που ασχολείται με ποινικέ υποθέσεις. Ε, μετανάστευση. Ε, είπατε ότι πέρυσι 200.000 Αφγανοί ε, προσπάθησαν, ε, έφτασαν στην Ένωση. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία αυτά είναι πολύ αξιόπιστα. Ίσως μπορούμε να έχουμε στο μέλλον πιο αξιόπιστα στοιχεία. Παρακαλώ, αν παρέλειψα κάτι, θυμίστε με. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Ντίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικά σχολεία και να απαντήσω. Ντανζόν. Δύσκολες ερωτήσεις, αλλά κέρυες δύσκολο να αποτιμήσει κανείς το ότι έχει πετύχει η αποστολή αυτή και εθνικέ δράσεις. Είναι δύσκολο να τα αποτιμήσουμε, ειλικρινά. Είναι πιο δύσκολο να αποτιμήσουμε το αντίστροφο, τι θα γινόταν αν δεν είχαμε πάει. Πάντως αυτά τα 9 χρόνια κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε επίπεδο μη εκτελεστικό. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε. Όσον αφορά υπουργεία, υπουργού, αστυνομικού κτλ. Προσπαθήσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα λογικής, όχι μόνο ευρωπαϊκό ή δικαιωμάτων, αλλά και κάποιες κοινέ διεθνείς αρχές. Παρά λοιπόν αυτά τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα, κάποιε φορές δεν γινόταν αυτό που λέγαμε. Είχαμε 9 υπουργού μόνο κατά τα τελευταία 9 χρόνια. Αρχίζαν από το μηδέν. Και αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είχε όψη Υπουργείου Εσωτερικών. Και την περίοδο 2007 με 9 σαν αρχηγείο στρατού και είχαν άλλη φιλοσοφία και οι προτεραιότητες. Και για την ISAF και την εκπαίδευση των αστυνομικών πρέπει να κατανοήσει κανείς τι μορφή θα έχει αυτή η αστυνομία πριν την εκπαίδευση. Γιατί βέβαια αυτή η αστυνομική δεν ήταν αστυνομική, ήταν στρατιώτες. Το ίδιο και αξιωματικοί. Τη αστυνομία. Οπότε, ίσως να μην ήμασταν όσο αποτελεσματικοί όσο θα έπρεπε. Και μετά οι μεταρρυθμίσεις και η υποστήριξη προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις σε επίπεδο νομοθεσίας νομοσχεδίων να υπάρχει τόσο πάντων εμπλοκή του αυγανικού στοιχείου με διακριτικά κλπ. Αλλά αυτά δεν έγιναν. Και αυτό ήταν απαγοητευτικό. Χωρίς πραγματική λοιπόν ηγεσία, όχι μόνο από τους παρατηρητές, αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν θα πρέπει να συνεχίσουμε. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι θα συνεχίσει την παρέμβασή της η Ένωση και μετά το 16, γιατί πρέπει να είμαστε παρόντες. Έχουμε θέματα όπως αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, σύνορα, μετανάστευση, τρομερά δικαιώματα που πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται να αφήσουμε τη δουλειά και ως Ευρωπαίος έτσι αισθάνομαι ότι έχω αυτή την ευθύνη. Η εντολή μας προέρχεται από τις χώρες μέλη. Είναι ευρύ αλλά και ταυτόχρονα περιοριστικό για το τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω ακριβώ ποια μορφή θα έχει η παρέμβασή μας μετά το Γενάρη. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα θέματα των γυναικών, αστυνομικών, ε, με τις ε, υπηρεσίες δίωξης, θα πρέπει να δούμε αν θα παραμείνουν αξιωματούχοι στις θέσεις τους. Πάντως, είχαμε πολύ καλή σχέση συνεργασία με άλλους διεθνείς εταίρους στην προσπάθειά μας αυτή και η αλήθεια είναι ότι στο Αφγανιστάν δεν λείπει η αρρωγή. Ούτε και τα χρήματα. Το θέμα είναι πώς δαπανώνται όλα αυτά και πώς εφαρμόζεται αυτή η αρρωγή γιατί από εκείνου νομίζω απορρέουν οι απογοητεύσει που ανέφερα προηγουμένω. Θα συνεχίσει πάντως τη δουλειά της μέχρι το τέλος εντολής η αποστολή, 31 του Δεκέμβρη, και θα προσπαθήσουμε μετά το Γενάρη να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε τουλάχιστον να μην χάσουμε, να μην απολέσουμε την καλή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για αυτή την συμβολή. Μήπως υπάρχουν άλλα μέλη που θα ήθελαν να προσθέσουν κάτι παρόλο που ήταν σύντομες αυτές τι παρουσιάσεις, ήταν ε, διεξοδικές. Και νομίζω ότι εκφράζω την πλειοψηφία των μελών που είναι υπέρ της συνέχισης της αποστολής. Βεβαίως συνεχίζει να αποτελεί ένα δύσκολο μέρος το Αφγανιστάν παρά τις συλλογικές μας προσπάθειες. Αλλά βεβαίως αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν ώστε να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα. Ευχαριστώ. Ε, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά με βάση αυτά που γνωρίζουμε σχετικά με το Αφγανιστάν και τον τρόπο που εξελίσσονται εκεί τα πράγματα, δεν ε, μπορούμε απλά να ε, χαιρόμαστε με τα όσα έχουν γίνει, αλλά να θέσουμε στο Συμβούλιο το θέμα της ανανέωσης των αποστολών μας στο Αφγανιστάν. Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορεί να κάνει η Γιούπολ Ίσως θα έπρεπε να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο. Ε, ε, υποστήριξη προς τις αστυνομικές δυνάμεις ή προς, τον, ή προς τις ε, ένοπλες δυνάμεις στο στρατό ή υποστήριξη για την ε, καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Αλλά από αυτά που ακούμε νομίζω ότι έχουμε σπαταλήσει χρήματα, κόπο, χρόνο Μα συγγνώμη, αυτό είναι ο, ο, λόγος που, που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους για να σκεφτούν, για να σκέφτονται τι ακριβώς μπορούν να κάνουν και σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο ειλικρινείς ε, για τα όσα συμβαίνουν. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι γελίο αυτό που συμβαίνει. Πρόκειται για κατασπατάληση των ε, χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων και μάλιστα χωρίς να επιφέρουμε και κανένα θετικό αποτέλεσμα για τους Αφγανούς. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, βέβαια δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο εκφοράς με την Άννα. Εκείνη ε, είναι λίγο πιο έντονη ίσω από μένα. Εγώ συμμερίζομαι όμως την ε, διαπίστωσή της. σα ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσία σα εδώ, για αυτήν την παρουσίαση και για την ειλικρίνειά σα, Αλλά μου επιβεβαιώνει την αντίληψη που ομολογώ ότι είχα ήδη διαμορφώσει μετά από τι επισκέψει μου και συζητήσει. Επιβεβαιώνει λοιπόν την αντίληψή μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα για τέτοιες αποστολές. Αλλάζει η κατάσταση στο Αφγανιστάν, αλλάζει η κατάσταση στην Ένωση. Συμμερίζομαι αυτό που είπε ο κύριος Ντίν. Όντως πρέπει να θέτουμε θέματα αποτελεσματικότητας, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και προσέγγιση ε, ίσως υπάρχει, είμαι πεπισμένος μάλιστα ότι υπάρχει χρησιμότητα. Αν δεν ήμασταν εκεί θα ήταν χειρότερη κατάσταση, αλλά με τι τρόπο ε, η μη στρατιωτική αποστολή που έχουμε εδώ και 9 χρόνια, μην ξεχνάμε 9 χρόνια, έχει έννοια, μήπως χρειάζεται περισσότερο στρατιωτική παρέμβαση. Προσωπικά δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τέτοιο ρόλο σήμερα στο Αφγανιστάν. Πρέπει να έχουμε μια αποστολή χώρο φυλακής που έχει αποδειχθεί χρήσιμη και αλλού. Μήπως ε, δεν θα έπρεπε να είναι μία αποστολή που να δίνει συμβουλές, θα μπορούσε να ήταν τμήμα της αντιπροσωπείας ε, της Ένωσης που δίνουν ε, μια και δίνουμε στρατηγικές συμβουλές στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν θα μπορούσαμε απλώς να διευρύνουμε την αντιπροσωπεία μας στην Καμπούλ για να έχουμε περισσότερες επαφές με το Υπουργείο Εσωτερικών ή Μήπως ε, θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με τη δικαιοσύνη και όχι με θέματα εσωτερικών. Είναι ερωτήματα απόλυτα πολιτικά, στρατηγικού χαρακτήρα. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε η Άννα Γκόμες. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά και το Συμβούλιο δεν πρέπει να αποφεύγει αυτά τα θέματα. Δεν θα πρέπει απλώς από χρόνο σε χρόνο να παρατείνει την εντολή χωρίς να εξετάσει πραγματικά σε βάθος τους λόγους ύπαρξής μας, παρουσίας μας στην Καμπούλ και με ποιο τρόπο θα έπρεπε να είμαστε παρόντες. Ωραία. Το σημειώνω. Και θα ζητήσουμε στους των πολιτικών ομάδων για το ποια μορφή θα έχει η επόμενη συνεδρίασή μας. Θα είναι σίγουρο ο κύριος Ντίν, αλλά θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την πολιτική συζήτηση για το τι χρειάζεται να γίνει στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πία Στένβολ για την παρουσίαση που έκανε σήμερα. Εγώ βλέπω ότι οι προσπάθειές της έχουν καρποφορήσει και η αστυνομική ακαδημία που συστάθηκε αποτελεί ένα πραγματικό επίτευγμα. Γι' αυτό θα ήθελα να την ευχαριστήσουμε για όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει μέσω της ε, Ιούπολ. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια χρονοθυρίδα μέσω της ε, γραμματείας μας για να βρούμε και χρόνο για να συνεδριάσουν οι συντονιστές και να δούμε πώς θα προχωρήσει ε, επί του θέματος αυτού η διαβούλευση και ελπίζουμε πριν από το καλοκαίρι να καταφέρουμε να παρακινήσουμε και το Συμβούλιο ώστε να λάβει αποφάσεις. Ωραία. Και με αυτό ολοκληρώνω την πρωινή μας συνεδρίαση. Σας καλώ να προσέλθετε στο εργαστήριο που θα διοργανώσουμε στις 3 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης και αύριο έχουμε εξαιρετικά σημαντικά θέματα στην ημερησία διάταξη. Παρακαλώ να είστε εδώ. Ευχαριστώ.